Okay, colleagues, I'm going to Να ας αρχίσουμε, συνάδελφοι. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε για το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Αν υπάρχουν προβλήματα από την κλέπω ευχαριστώ. Ανακοινώσει του Προέδρου. Να σα κάνω την επίσημη ενημέρωση από τη σύσκεψη των συντονιστών τη 30 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν πολλά, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Ε, έχουμε το πρόγραμμα για τις ακροάσει για τις αντιπροσωπείες. Ζητήσαμε από τις πολιτικές ομάδες να ενημερώσουν τη γραμματεία για τους προορισμούς που επιλέγουν για τι αντιπροσωπείες για το 2014. Μία επίσκεψη θα γίνει φυσικά για το πρώτο ημίση και το ίδιο για τις ε, δημόσιες ακροάσεις. Είχαμε επίσης την απόφαση των συντονιστών για την επιτροπολογία ε, και έλαβαν γνώση του ενημερωτικού δελτίου της 23ης Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα πεπραγμένα της συνεδρίας των συντονιστών της 30ης Σεπτεμβρίου, εντάξει. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Ουσιαστικά ένα σημείο έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Το πακέτο για τους σιδηροδρόμους. Ένα λεπτάκι να τα βάλω τα χαρτιά μου στη σειρά για να αρχίσουμε. Πρέπει να εγκρίνουμε πρώτα απ' όλα τα πρακτικά της συνεδρίας 16-17 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν προβλήματα, όχι ευχαριστώ. Το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους. Μέχρι τις 6 και 4 έχουμε χρόνο συνάδελφοι και θέλω να σας ενημερώσω ότι πρόκειται για την αρχική μόνο συζήτηση για αυτό το θέμα όπου μπορούμε θα έπρεπε να αποφύγουμε τις επαναλήψεις ε, των παρεμβάσεων των συναδέλφων ε, και στις προθέσεις μου ε, συγκαταλέγω ότι εξής. Πρώτον, σε σχέση με την έκθεση Ελκαντρέου με τους Σκιώδες, να ακούσουμε την παρουσίαση, να ακούσουμε την παρουσίαση του κυρίου Γκρόσε και του Σκιώδη, στη συνέχεια να ακούσουμε εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών και μετά εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη συνέχεια θα αφήσω χρόνο για τις ερωταπαντήσεις, τόσο ώστε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής να σχολιάσουν αμφότερες σημεία από τις δύο εκθέσεις και στη συνέχεια θα κάνω ακριβώς το ίδιο με την έκθεση Bilbao, Κράμερ και Ζιλ, Τσέλερ. και θα συνεχίσουμε με την, θα αφήσουμε την έκθεση Κόλιτσεκ προς το παρόν γιατί είναι εξίσου σημαντικό το θέμα αλλά δεν είναι εισάρθμες οι τροπολογίες. Ε, γι' αυτό επιλέγουμε αυτή τη σειρά. Ε, Σα παρακαλώ να με βοηθήσετε για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Θα έχουμε τέσσερα λεπτά για τους εισηγητές 3 λεπτά για τους κοιόδη, Επιτροπή των Περιφερειών. Ένα πεντάλεπτο. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ένα πεντάλεπτο για τις δύο πρώτες, για ένα πεντάλεπτο για τις τρεις επόμενες και δύο λεπτά για την έκθεση Κόλιτσεκ. Ε, και όλοι οι υπόλοιποι έχουν δύο λεπτά έκαστος. Με αυτά ευελπιστώ ότι θα τηρηθεί το διαγραμμα. Αρχίζουμε με τον ε, Σαΐντελ Αντράουι. Ε, και μην το πάρετε προσωπικά, αλλά θα βάλω και χρονόμετρο. Ε, ε, Ελχαντράουι, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, είναι μια μεγάλη τιμή για μένα που παίρνω πρώτο το λόγο διότι εγώ έλαβα τις περισσότερες τροπολογίες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας θυμίσω ε, ποιο είναι το πνεύμα που διαπνέει την ε, έκθεση μου θα ήθελα να σας πω ότι η απελευθέρωση της αγοράς δεν μπορεί να συνιστά αυτό σκοπό επουδενή. Του τουλεχθέντος μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για να υπερπηδήσουμε τα οικονομικά εμπόδια και να τονώσουμε την οικονομική μεγέθυνση. Αυτό θα το επιτύχουμε μόνο αν ταυτόχρονα με το άνομα της αγοράς ενισχύσουμε και την κοινωνική προστασία των εργαζομένων και μια πιο ε, αυστηρότερη ε, ρύθμιση σε σχέση με την ενημέρωση των ταξιδιωτών, σύστημα τιμολόγησης, σε νέο σύστημα έκδοση εισιτηρίων. Χρειαζόμαστε επίση και ισορροπία ανάμεσα στην παροχή δημόσια υπηρεσία και το άνοιγμα ε, τη αγορά. Ε, Επιλογέ αλακάρτ λοιπόν που θα κληθούν να κάνουν ε, όλοι. Χρειάζεται να κατοχυρώσουμε μια ευελιξία και ένα δίκτυο χάρη στο οποίο θα έχουμε ένα μίξ δημοσίων υπηρεσιών ανοιχτών για το κοινό την κατοχήρωση για τους ε, επιβάτες μιας ομοιομορφίας υπηρεσίας ε, δεδομένης και της ετερομοιομορφίας ε, σε ετερομορφία συγγνώμη, ως προς τις υποδομές, τα συστήματα, τα υποσυστήματα που χρησιμοποιούνται. Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα ενημερώνονται σωστά οι καταναλωτέ για να υποφεληθούν από αυτήν την νέα κατάσταση. Ως προς τις υποδομές, στο μέτρο που υπάρχουν ελεγκτικές αρχές, εθνικές ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να ενισχυθούν, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να λάβουμε υπόψη την περίπτωση των κάθε ολοκληρωμένων επιχειρήσεων. Σχετικά έχω καταθέσει και διάφορες τροπολογίες. Έχουμε 540 τροπολογίες, 540 για την έκθεσή μου και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Έχω προαναφερθεί σε αυτά. Κάποιοι μίλησαν για την υποδομή, για το άνοιγμα της αγοράς την ισορροπία που πρέπει να επιτύχουμε επιμέρους διατάξεις που σχετίζονται με τα δίκτυα μεταφορών, έκδοση εισιτηρίων, διαχείριση υποδομών, επιτροπές συντονισμού που πρέπει να συγκροτηθούν, πώς θα χρησιμοποιηθούν, ποιος θα είναι ο ρόλος της Εθνικής Αρμόδιας Ελεγκτικής Αρχής και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ε, θα ήταν καλό να αποφύγουμε οποιοδήποτε δόγμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να υιοθετήσουμε ανταυτού ε, μια επικοδομητική προσέγγιση. Έχουμε ήδη κάνει διάφορε συσκέψει με του κοιότητες εισηγητές. Έχουμε προβλέψει μελλοντικά διάφορε συνεδριάσει με τρόπο ώστε μέχρι το τέλο του τρέχοντος να ικανοποιηθούν όλοι στο μέτρο του δυνατό από το αποτέλεσμα. Έχουν καταδεχθεί διάφορες τροπολογίε για τα συστήματα. Ε, το άρθρο 7 είναι μια προτεραιότητα για μεγάλο αριθμό μελών της Επιτροπής και ε, κάποιοι ε, συμφωνούν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιλέγουν την οδό της αναθεώρησης. Υπάρχουν άλλες τροπολογίες που επιθυμούν περισσότερα, θέλουν να υπερβούν και να συμπληρώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε σχέση με το άνοιγμα της αγοράς ε, έχουν αναφερθεί διάφορα σημεία. Υπάρχει το φάκελος PSO παραδείγματος χάρη, η αμοιβαιότητα, η διαλειτουργικότητα, διάφορες ε, τροπολογίες που σχετίζονται με την τιμολόγηση και την έκδοση εισιτηρίων και από ό,τι φαίνεται ε, έχει εξευρεθεί ε, μία συμβαστική λύση χωρίς να έχει επισημοποιηθεί ακόμη. Τέλος πάντων θα περιοριστώ σε αυτά τα σχόλια εν κατακλείδη να ε, τονίσω ότι με άκνες προσπάθειες θα κάνω ό,τι πένα από το χέρι μου για να καταλήξουμε σε μία κοινή, κοινώς αποδεκτή λύση. Ευχαριστώ κύριο Καντσιάν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Αλκαντράουι για τα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Στις συνεδριάσεις ε, που κάναμε από κοινού θεωρώ ότι καταφέραμε να διευκρινίσουμε λίγο τις απόψεις των μεν και των δε. Ε, εγώ ξεκινώ από την προϋπόθεση ότι η βασική αρχή είναι το άνοιγμα των αγορών για όλα αυτά. Διότι αν δεν υπάρχει άνοιγμα στις αγορές, νομίζω ότι αρκετά από αυτά τα οποία συζητούμε εδώ δεν ε, έχουν κανένα νόημα. Υπάρχουν κάποιες ενθαρρυντικές τροπολογίες από αυτά που διάβασα, διότι είδα τις μεταφράσεις σήμερα το πρωί, οπότε δεν μπόρεσα να επισέλθω σε λεπτομέρειες για τις τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι μπορώ να θεωρήσω ότι αρκετές τροπολογίες υποστηρίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιβεβαιώνουν και ενισχύουν την απελευθέρωση των αγορών σε τοπικό επίπεδο, τα βελτίωση για τους επιβάτες για να μπορέσουμε να έχουμε μια ενιαία σιδηροδρομική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η βασική μας αρχή. Ελπίζουμε λοιπόν να μην διακυβεύσει κανείς αυτή την αρχή με μια σειρά από παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις που θα επιτρέψουν να ερμηνεύει ο καθένας σε εθνικό επίπεδο αμφίσιμους κανόνες. Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι ότι πριν φτάσουμε στη διακυβέρνηση θα πρέπει να υπάρχει ένας εθνικός ρυθμιστής και ένας ευρωπαίος ρυθμιστής. Κατά την άποψή μου είναι και οι δύο ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να επιτύχουμε τη διακυβέρνηση η οποία δεν θεωρώ ότι θα πρέπει από αυτά που είδα από αρκετούς συναδέλφους ε, να θεωρήσουμε ότι την ε, περιχαρακώνει το συνικό τείχος ε, ή υπάρχει μια πλήρης απελευθέρωση, αλλά θα υπάρχουν μια σειρά από κανόνες που θα επιτρέπουν μια χωρίς διάκριση πρόσβαση στο δίκτυο και ταυτόχρονα θα επιτρέπουν να υπάρχουν και απαραίτητε συνέργειες για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα τομέα όπως είναι αυτός των σιδηροδρόμων τόσο περίπλοκο. Θεωρώ λοιπόν ότι η δυνατότητα να έχουμε πλήρες άνοιγμα των αγορών, να έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρυθμιστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μαζί με το εθνικό δίκτυο ε, ρυθμιστών θα καταφέρουμε να ρυθμίσουμε αυτές τις σημαντικές πτυχές ε, τις οποίες έχουμε αναφέρει και υπάρχει και σχετική μου τροπολογία θεωρώ ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ρύθμιση και ως προς το κόστος και όσον αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά. Όσον αφορά τη διάθεση των εισιτηρίων, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει να μην γίνονται συμφωνίες καρτέλ που θα κάνουν οι διάφοροι διαχειριστές των συστημάτων, διότι έτσι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματική ανταγωνιστικότητα, αλλά να έχουμε ένα πραγματικά ενιαίο εισιτήριο ε, που θα είναι ένα τοπικό εισιτήριο ε, συν ε, οποιαδήποτε, για πολλούς ε, άξονες σιδηροδρομικούς και ταυτόχρονα να μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιήσει. Έτσι να μπορούμε να έχουμε προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστούμε κύριε Καντσιάν. Ξέρω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα, αλλά μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Ντιμπάκερ για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες προς και κατά την άποψή μου υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες αποδυναμώνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άποψή μου έκανε μια πρόταση που μας προσδίδει τη δέουσα ισορροπία από την οποία θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Εμείς έχουμε εκφράσει την άποψή μας ε, πριν από κάποιες εβδομάδες για αυτή την αναδιατύπωση και τώρα πλέον δεν θα πρέπει να απομακρυνθούμε τόσο πολύ από αυτά στα οποία έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν εδώ κάποια σημαντικά ζητήματα. Καταρχάς το θέμα της διακυβέρνησης, της governance. Η άποψη της πολιτικής μας ομάδας για τη διακυβέρνηση είναι ότι προκειμένου να ανοίξει η αγορά θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε δυνατότητες ε, να έχουμε ίσους όρους ε, για τις υποδομές αλλά και για τους διαχειριστές του δικτύου. Επομένως το unbundling είναι ο κατάλληλος τρόπος για να καταλήξουμε στον ε, σε αυτό που επιθυμούμε. Αυτό όμως δεν είναι τόσο εύκολο στο Κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει αρκετή πλειοψηφία κατά την άποψή μου. Αναφερθήκαμε σε οικονομικές λύσεις σε διάφορα σημεία. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το συνικό τείχος εάν δεν υπάρξει δυνατότητα απελευθέρωσης ε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να καταλήξει σε πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το συνικό τείχο λοιπόν το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονομική ροή δεν ξέρω αν μπορεί να επιτευχθεί ή αν μπορούμε να το ενισχύσουμε περαιτέρω. Υπάρχει και το θέμα του ανοίγματο των αγορών για του επιβάτε σε εθνικό επίπεδο, του εγχώριου. Αναφερθήκαμε στο θέμα της ε, αλλαγής των ε, διαφορών δικτύων. Το άνοιγμα της αγοράς έχει βελτιώσει τον ανταγωνισμό, θα πρέπει να τον βελτιώσει περαιτέρω και θα πρέπει όμως να βελτιωθεί και η ποιότητα προς όφελος των επιβατών. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σαφή θέση για το θέμα αυτό. Κατόπιν, το θέμα της οικονομικής ισορροπίας. Ε, καταθέσαμε σχετικές ε, τροπολογίες ώστε οι υπηρεσίες που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, οι ε, υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης, να παραμείνουν και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό για να κλείσει οριστικά η αγορά και να μην υπάρχει πρόσβαση για άλλους. Πρέπει να σκεφτούμε και υπό το πρίσμα των πελατών. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα εισιτήρια και θα πρέπει να κάνουμε και μία απόπειρα να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση σε αυτό το σημείο ο ανεξάρτητος ε, ρυθμιστής σαφώς και είναι σημαντικός. Δεν μπορούμε να αφήσουμε πάσα ελευθερία στο κράτος μέλος για να ε, ρυθμίζει τα πάντα ε, κατά το δοκούν και να αποδυναμώσει ουσιαστικά τους κανόνες. Πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση, δεν θα είναι εύκολο και δεν θα είναι εύκολο να καταλήξουμε σε συμπερασμό. Ευχαριστώ κύριε Ντιμπάκερ. Να καλωσορίσω κάποιους επισκέπτες του κυρίου Λάιχτριντ από την Αυστρία και έχουμε και κάποιους πράσινους ακτιβιστές ε, από τον κύριο Ζαρίμπη. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν όλους εδώ σήμερα. Η κυρία Ντουράν θα μιλήσει για τρία λεπτά εκ μέρους του κυρίου Μπίσερ. Ευχαριστώ και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που αποδεχόμαστε, είναι κοινέ. Υπάρχουν τρία σημεία που θα ήθελα να τονίσω αντίθετα. Πρώτον, σε σχέση με τις υπέρμετρα μεγάλες αρμοδιότητες που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους διαχειριστές υποδομών στο μέτρο που θέλει να καταργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εφιστάμενη δυνατότητα να ανατεθεί σε εξωτερικό ανεξάρτητο οργανισμό η τιμολόγηση και η έκδοση των εισιτηρίων ναι, κέρια σημασία σε αυτές οι υπηρεσίες και ε, ε, έχει θεμελιώδη σημασία να αποφύγουμε τις καταχρήσεις αυτού του ε, μελλοντικού μονοπωλίου των διαχειριστών υποδομών. Δεύτερο σημείο, μη διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τους παρόχους ως προς την πρόσβαση στο δίκτυο πρέπει να εξακριβώνεται και να εγγυείται από μια κρατέα ρυθμιστική αρχή αυτή η πρόσβαση. Όμως ταυτόχρονα δεν χρειάζεται οι διαχειριστές υποδομών και οι φορείς, η παροχή να διαχωρίζονται πλήρως στο μέτρο που ανήκουν στον ίδιο ενοποιημένο όμιλο. Ε, ε, το έχω επαναλάβει στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι προκρίνει αυτό το σύστημα, το οποίο όμως συνεπάγεται επιπρόσθετο κόστος ε, διαφορά προ προς τους στόχους που διαταράζει τη συνοχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος και συνιστά διακριτική μεταχείριση. Τρίτον, σε σχέση με τη μελλοντική χρηματοδότηση και την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, βλέπουμε σήμερα τι έχει συμβεί στον τομέα των, εμπορευμάτων, των εμπορευματικών μεταφορών. Ε, η απάντηση λοιπόν είναι δικλείδες ασφαλείας, ούτως ώστε στον τομέα δημοσίων υπηρεσιών να μην επιδιώκουμε μόνο τη χαμηλότερη τιμή, αλλά και ικανοποιητική ε, ποιότητα ε, υπηρεσιών για το ticketing, την έκδοση εισιτηρίων. Σας το ξαναείπα στην αρχή της παρέμβασής μου, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, κυρίως να έχουμε ένα δυσυνοριακά λειτουργό σύστημα. Ευχαριστούμε. Κύριε Βλάσσα είστε έτοιμος γιατί Βλάσακα από συντηρητικού, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τσεχικά, την μητρική μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ και τον εισηγητή για την πρόταση που κάνει, για τα συμπεράσματά του. Εγώ υποστηρίζω την ε, διεύρυνση του συστήματος ε, για τα εισιτήρια είναι όντως ε, σημαντική συμβολή για τους πελάτες των δικτύων. Ξέρω βεβαίως ότι αυτό το σύστημα για να διαμορφωθεί θα είναι μεγάλη πρόκληση. Και θα ήθελα να σας τονίσω το εξής. Για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια ε, θα γίνει την Τετάρτη μια εκδήλωση στις 10. Ε, αν δούμε τις ε, τροπολογίες βλέπουμε ότι από τις μελισσότερες ομάδες μιλούμε για διαχωρισμό των υποδομών από τις εταιρείε. Εγώ υποστηρίζω τις τροπολογίες οι οποίες θέλουν να εξασφαλίσουν ίσες προϋποθέσεις για την επιλογή μεταξύ των εταιριών ή ενός ξεχωριστού μοντέλου. Αλλά ε, όλες τις τροπολογίες που επιβάλλουν περιορισμούς ε, σε ό,τι αφορά την, η μετάβαση από το ένα στο άλλο μοντέλο ε, δεν μπορώ να τις δεχτώ. Ε, επίσης, αυτό το διτό χαρακτήρα των ε, ε, προτάσεων πρέπει να τον επικροτήσουμε. Οι εταιρείε, βέβαια, ίσως να δημιουργήσουν διακριτική μεταχείριση και σε άλλους τομείς, πέραν των σιδηροδρομικών μεταφορών, σε άλλου τομεί που ίσω δεν έχει αναφέρει η Κομισιόν. Για παράδειγμα, για την μισθοδοσία των υπαλλήλων. Και ένα τελευταίο τομέα είναι η εκπροσώπηση ε, των ε, ε, υπηρεσιών και όσων παρέχουν τις υπηρεσίες στους σιδηροδρόμους στις όλες τις διαπραγματεύσεις. Εδώ μιλούμε για τη διαφάνεια των τιμών και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αν ε, ε, οι σιδηρόδρομοι θέλουμε να είναι ένα ε, μέσο ποιοτικό και που μπορεί να το πληρώσει ο κόσμος για να το χρησιμοποιήσει σε σχέση με την οδική, τις οδικές μεταφορές, θα είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Wills, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Η δική μου ομάδα από την αρχή είχε, υποβάλει, είχε αναφέρει την κριτική της ε, ε, στο πακέτο αυτό και είναι η μόνη που είχε βάλει ε, τροπολογίες για καταψήφιση αυτής της πρότασης. Μιλούμε για διαρθρωτικές απαιτήσει, όπως την οδηγία για την αναδιατύπωση που διευκολύνουν περισσότερα μοντέλα διακυβέρνησης. Η πρόταση της Κομισιόν θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαχωρισμού που εμείς θεωρούμε ότι είναι και κίνδυνος αλλά και διακριτική μεταχείριση για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί επιτροπολογίας. Όπως και στις τροπολογίες μας έχουμε αναφέρει, είμαστε υπέρ της διατήρησης των δυνατοτήτων ενός ολοκληρωμένου συστήματος που μέχρι τώρα υπάρχει, που προσφέρει ε, ισορροπία, που δεν διακυβεύει ε, τον πλουραλισμό των ε, συμμετεχόντων στις μεταφορές, και που μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπει το διαχωρισμό ε, ε, των υποδομών από τις ε, εταιρείε. Από την δική μας λοιπόν προσέγγιση απορρέει ότι δεν είμαστε συμφωνοί με την άποψη του ΕΛΚ και άλλων ομάδων που μιλούν για πλήρη διαχωρισμό και τον θεωρούν αυτό ως μοναδική εναλλακτική και αποκλείουν οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για τους σιδηροδρόμους. Αυτά που αναφέρονται στο 7α, 7β και 7γ από την Κομισιόν, το μοντέλο που αναφέρεται στα άρθρα αυτά, για το συνικό τείχος θα συμβάλλει ώστε να υπάρξει προσθέμενη αξία για τους σιδηροδρόμους. Για την 43 του 2012 οι προθυποθέσεις ήδη υπάρχουν και δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Ε, είναι θετικό βέβαια ότι και άλλοι εκπρόσ... Ε, ε, ευρωβουλευτές και από, το... από τους σοσιαλιστές και από άλλες ομάδες δείχνουν ότι αυτές οι τροπολογίες που αναφέρουν διαγραφή τμήματων των προτάσεων της Κομισιόν τις υποστηρίζουν. Αυτό καθιστά σαφές ότι πολλές πτυχές του κειμένου ή και το σύνολο του κειμένου ε, δεν είναι ε, απαραίτητο και θα πρέπει να διατηρήσουμε το status quo. Και τέλος μια παρατήρηση για τη συζήτηση για, τον, ε, για τη ρυθμιστική αρχή. Σημαντικό είναι για μας να πούμε ότι μια τεχνική εντολή θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν διαιτητή και δεν θα πρέπει να υπάρχει πολιτική χρειά σε αυτόν τον ενδιάμεσο που θα παρέμβει. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Βίλς. Ο κύριος Μαγκάν τώρα από την Επιτροπή των Περιφερειών να μας πει την άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών. Ε, υποθέτω θα μας δώσετε την άποψή σας για όλο το πακέτο, οπότε παρακαλώ, έχετε το λόγο. Euh, ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Ε, θα ήθελα να σας μιλήσω εν ολίγης για την γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών που θα είναι σε λίγο διαθέσιμη και στη δική σας ιστοσελίδα την οποία εμείς εγκρίναμε ε, πριν από λίγες ημέρες στην Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών. Θέλω να σας πω ότι εγώ ήμουν ο μοναδικός συγητής στην Επιτροπή των Περιφερειών. Εδώ υπάρχουν έξι συγητές από ό,τι κατάλαβα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να επικεντρωθώ σε αυτά που έκρινα εγώ πιο σημαντικά, πιο απαραίτητα ως προς ε, τις ε, αρχές που την τοπική κυκλοφορία. Ε, ρίξαμε το βάρος λοιπόν στην εκπροσώπηση αυτών των τοπικών εταιριών στα διάφορα όργανα διακυβέρνησης, ε, κυρίως ε, ως προς τους διαχειριστές ε, των υποδομών. Γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι συχνά οι διαχειριστές υποδομών χρησιμοποιούν τοπικές υποδομές που συχνά χρηματοδοτούνται από ΟΤΑ, από αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε θεωρούμε ότι είναι λογικό στα πλαίσια τη διακυβέρνηση να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση αυτών των αροχών. Επίση, ε, επιμείναμε στη σημασία των επιχειρηματικών σχεδίων μεταφορών. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι πραγματικά προγράμματα που θα προαγάγουν την διατροπικότητα, τη διασυνδεσιμότητα και θα προστατεύουν τις μεθοριακές κυρίως περιοχές. Εγώ είμαι αλσάτος και αντιλαμβάνομαι πόσο επικίνδυνο είναι ένα ε, επιχειρηματικό πρόγραμμα που καλύπτει μόνο τη δική μου περιοχή και όχι την παρακείμενη περιοχή μετά τη διέλευση των συνόρων ενώ η ίδια τοπική κατάσταση επικρατεί και στις δύο περιοχές ε, εξού και σημασία των, ε, της καλής διασυνοριακής συνεργασίας για τις μεθοριακές περιοχές περιοχές. Επίσης, ασχοληθήκαμε με τη διευκόλυνση των ε, διαχειριστών, κυρίως όταν υπάρχει αλλαγή διαχειριστή ε, υποδομής. Εμείς δεν επιλέξαμε για την ε, άμεση ανάθεση ή για την, τους διαγωνισμούς. Πιστεύουμε ότι η επιλογή θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση από τη ρυθμιστική αρχή. Η ρυθμιστική αρχή πρέπει να εκδίδει γνωμοδότηση εάν η τοπική αρχή καταγγέλει την άμεση ανάθεση εντοπίζοντας ε, το, ως πρόβλημα το ζήτημα των κριτηρίων. Τώρα, ε, ποια είναι η αξία του τροχαίου υλικού και τι μισή της ε, δεν θα έπρεπε σε, μεταφορά, σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή υποδομής να δημιουργείται πρόβλημα λόγω της αξιολόγησης του τροχαίου υλικού. Επίσης για τα διασυνοριακά προγράμματα η χρηματοδότηση δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ε, αμοιβαία χρήση ε, του τροχαίου υλικού, διασυνοριακή χρήση του τροχαίου υλικού. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια εναλλακτική λύση. Σε το επικό επίπεδο και πάλι θα θέλαμε να σπεράσουμε περάσουμε κάποια συγκεκριμένα μηνύματα για τη διακυβέρνηση. Εάν έχουμε το κάθετα ολοκληρωμένο μοντέλο ή το χωριστό μοντέλο θα είναι μια επιλογή των κρατών μελών, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε απόλυτη ε, χρηματοοικονομική διαφάνεια και πλήρη ανεξαρτησία του διαχειριστή. Και γι' αυτό επιλέγουμε να υιοθετηθεί η πρόταση, αυτό ε, προτείνουμε μέσα στη γνωμοδότησή μας. Ε, τώρα, η βασική της των σιδηροδρομικών υπηρεσιών θα πρέπει να μετέχουν στην διαδικασία επιλογής και ανάπτυξη των υπηρεσιών. Επίσης, η συνεργασία ανάμεσα στους διαχειριστές υποδομών είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να προωθήσουμε τις διασυνοριακές συνδέσεις που έχουν τόσο μεγάλη βαρύτητα για κάποιες περιοχές για το θέμα λοιπόν αυτό η Επιτροπή των Περιφερειών κρίνει ότι ε, με την συγκρότηση του δικτύου των διαχειριστών υποδομών δυνάμει της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε μια νέα ευκαιρία που ανοίγεται μπροστά μας για να καλύψουμε τις τοπικές ανάγκες. Ε, οι τοπικές ε, ρυθμιστικές αρχές σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσουν πρόσκομα στην προώθηση της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 διαλειτουργικής ε, μεταφοράς ε, επιβατών, είτε μιλάμε για τη μακροκλίμακα, εξετάζουμε το θέμα των μεταφορών δηλαδή σε ευρωπαϊκή κλίμακα, είτε το εξετάζουμε υπό το τοπικό πρίσμα. Θεωρώ ότι αυτοί οι κανόνες ε, που τώρα θεσπίζουμε θα πρέπει να εφαρμόζονται από έναν ισχυρό, ανεξάρτητο και διαφανή ρυθμιστικό φορέα. Φυσικά ο ρυθμιστικός φορέας δεν θα καθορίζει τους κανόνες ε, θα παρατηρεί και θα εποπτεύει την εφαρμογή τους. Η νομοθεσία αυτή μπορεί να λειτουργήσει μόνο υπό τρεις προϋποθέσεις. Η ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ισχυρή, να έχει τα χρηματοοικονομικά και άλλα μέσα για να δράσει και από ό,τι φαίνεται στη χώρα μου τουλάχιστον δεν επιλέγεται αυτή οδός προς το παρόν. Δεύτερον πρέπει να είναι επαρκής ε, ο φορέας ούτως ώστε να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες δεξιότητες, να καλύπτει τις απαιτήσει που θέτουμε για τις ρυθμιστικές αρχές και μην ξεχνάμε και τον απότερο στόχο της μεταρρύθμισης να είναι πιο ελκυστικές οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Ε, δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα νέο καθεδρικό ναό ή να ε, τραγουδήσουμε μία οδή στην απορρίθμιση. Ο στόχος μας είναι να ε, είναι ο ελκυστικότερος ο τομέας ε, των μεταφορών για τους επιβάτες και ξαναλέω ότι εκπροσωπούμε και ασχολούμαστε εδώ ε, με τις απόψεις των τοπικών ρυθμιστικών αρχών που αν δεν εμπλακούν επαρκώς στον προσδιορισμό της νέας αρχιτεκτονικής διακυβέρνησης δεν θα μπορείς να κατοχυρωθεί η ποιότητα των νέων υπηρεσιών. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, και ελπίζω να προλάβετε να πάρετε ε, το τρένο για να γυρίσετε στην Αλσατία και εμείς τα ξέρουμε αυτά γιατί παίρνουμε συνέχεια το τρένο και πηγαίνω ερχόμαστε όπως ξέρετε. Έχουμε τον κύριο Κράμερ, Ιλκέ και Ρότερ. Ποιος άλλος θέλει το λόγο για, για την έκθεση αλκαντράου έτσι. Δύο λεπτά έκαστος και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κράμερ, δύο λεπτά. Μάικλ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Όντως ε, πρέπει να προχωρήσουμε με ρεαλιστικό τρόπο, να μην ε, κάνουμε επιλογές από το ένα ή το άλλο σύστημα. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα καλό σύστημα, αλλά στην Γερμανία ας πούμε υπάρχει ένας ε, ε, κλαδικός, ε, μια κλαδική τιμή, ένα τιμολόγιο και στη δική μου τη χώρα επίσης υπάρχουν ελάχιστοι μισθοί και για εκεί υπάρχει, υπάρχουν προβλήματα με το κοινωνικό ντάμπινγκ, αλλά έχουμε θετικές εμπειρίες γιατί έχουμε την μεταφορά των αγαθών και δεν ξέρω καμία χώρα όπου οι αγορά της, το άνοιγμα της αγοράς για την μεταφορά αγαθών είχε αρνητικά συνέπειες. Είχε παντού θετικές συνέπειες, αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης ε, που υπήρξαν σε πολλές ε, χώρες και θα πρέπει να τα καταφέρουμε και εμείς. Ε, η ανεξάρτητη τώρα αριθμιστική αρχή βεβαίως είναι αποφασιστική σημασίας και ε, έχω, δίνω δίκιο στον ε, ομιλητή που μόλις πήρε το λόγο. Ε, πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και να την αποδυναμώσουμε είναι ο λάθος δρόμος. Τώρα για την ροή των μετρητών θα πρέπει να προσέξουμε. Εμείς δεν θέλουμε να καταβαρωθρωθεί η διαφάνεια. Ούτε θέλουμε ε, να αγοράζει η μία εταιρεία την άλλη και να, γίνει, να καταλήξουμε τελικά σε ολιγοπόλια ή μονοπόλια. Ε, το τελευταίο σημείο, που το είπε και, ο, ε, και η κυρία Βίλμς, ε, πρέπει να, να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τους σιδηροδρόμους. Θα πρέπει όμως αυτό να μην γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί δεν γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η, το γερμανικά τρένα πάνε στο, στα ολλανδικά, ας πούμε, στους ολλανδικούς σιδηροδρόμους, χωρίς όμως να τους ανήκουν οι ράγες των τρένων τα, το ποσοστική σημασία είναι άλλο πράγμα και όχι αν θα υπάρξει διαχωρισμός α, της παροχής υπηρεσιών ή των δικτύων. Εμείς θέλουμε να υπάρξει διαχωρισμός λοιπόν μεταξύ των α, δικτύων και των υποδομών. Ο κύριε... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον Σαΐτ για την έκθεσή του, η οποία είναι πολύ ισορροπημένη. Θα ήθελα, χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, να σταθώ σε δύο θέματα. Υπάρχει ε, το θέμα της υποδομής, ε, το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εγώ εξακολουθώ να είμαι υπέρ της απόλυτα ξεχωριστής υποδομής, που ήταν η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι οι μεγάλοι σιδηροδρομικοί φορείς που έχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες έχουν ε, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους ε, παροχής ε, υπηρεσιών. Θα πρέπει να βασίζονται οι όροι στην ισότητα της πρόσβασης της αγοράς, ισότητα της πρόσβασης στις υποδομές και αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα στην πραγματικότητα είναι το μόνο θετικό στοιχείο. Το να έχουμε πλήρη διαχωρισμό θα ήταν το πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση. Το δεύτερο σημείο, το οποίο θα ήθελα να πω, είναι πιο συγκεκριμένο για τα θέματα της, της έκδοσης εσωτερίου, στο οποίο αναφέρθηκε και ο εισηγητής. Ε, είναι πραγματικά κίνδυνος ε, να βλέπουμε τι γίνεται με τους παρόχους ε, που θα φτάσουν απευθείας στις εμπορικές πολιτικές για τους σιδηροδρόμους. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό σε επίπεδο πληροφορικής και λογισμικού, αλλά να είναι καταστροφικό για τους σιδηροδρόμους, διότι δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Ε, σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι η έκθεση είναι αρκετά ισορροπημένη και ε, πρέπει να βρούμε τι γίνεται με την ανοιχτή πρόσβαση και τη σύμβαση ε, παροχή των υπηρεσιών, ε, την απευθείας ανάθεση, όλα αυτά τα θέματα. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι τελείως ε, διαφορετικά και θα πρέπει να τα προσέξουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέρτοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω εγώ τον εισηγητή. Όντω δεν είναι πολύ εύκολο να τοποθετηθεί κανεί για αυτό το δύσκολο και αρκετά συναισθηματικό θέμα. Νομίζω ότι η γενική θέση ε, θα πρέπει να είναι υπέρ μιας ισόρροπης προσέγγισης ε, για την ε, συζήτηση αυτή για, την, για το διαχωρισμό των δύο επιλογών. Δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε με ακραίους τρόπους και να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό και αυτή την διαδικασία ήδη την έχουμε δει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου μέσω και της αναδιατύπωσης και τα καθήκοντα που θέσαμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να ενισχύσουμε τις ρυθμιστικές αρχές. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, ροή των ε, κονδυλίων, βεβαίω είναι σαφέ ότι τα χρήματα δεν μπορούμε να τα καταχρώμεθα, αλλά σε αυτή την αναδιατύπωση έχουμε μια πολύ ευρεία ενίσχυση της αριθμιστική αρχή. Ε, σε ό,τι αφορά την, ε, την, υποχρέωση ε, ενημέρωσης και διαφάνειας, έχουμε πάει αρκετά μακριά, θα μπορούσαμε να πάμε και πιο μακριά. βέβαια η πρόταση της δεν μπορούσαμε να περιμένουμε την πρόταση Κομισιόν μέχρι να εφαρμοστεί η νομοθεσία της στα κρατημέλη και τώρα έχουμε το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους και θα θέλαμε ε, λόγω αυτής της συζήτησης αυτού αυτούς τους σημαντικούς φακέλους ας μην τους αφήσουμε στις ε, καλένδες για τους τεχνικούς φακέλους μιλώ εγώ κυρίως. Είμαι της άποψης ότι αν δεν προχωρήσουμε καταρχάς Ας ε, ε, αφήσουμε αυτό τον ε, φάκελο στην άκρη, να δούμε τα τεχνικά του ζητήματος, τα τεχνικά σημεία και επίσης νομίζω ότι εδώ στις Βρυξέλλες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε το θέμα της επικουρικότητας γιατί Έχουμε πολλά αποτελέσματα από, πολλές από ε, ε, πολλά κράτη-μέλη όπου ε, βλέπουμε τι γίνεται με τα διάφορα ακροδεξιά κόμματα κτλ. Ας είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί, ας μην διαχωρίσουμε τις υποδομές από τις παροχές και ας αφήσουμε, αν είναι να προχωρήσουμε σε κάτι, να προχωρήσουμε στα τεχνικά θέματα. Να καλωσορίσουμε άλλο ένα γκρουπ από την... Ε, Αυστρία, αν θέλετε να καθίσετε, όπου βλέπετε πράσινο καρτελάκι μπορείτε να καθίσετε στις θέσεις των αναπληρωματικών μελών. Αλλά τώρα δεν γίνεται να στέκεστε, αφόσον υπάρχουν θέσεις, καθίστε. Λοιπόν, ο κύριος Φρυγκόλ για δύο λεπτά. Ναι, συμφωνώ και εγώ με τις παρατηρήσεις του Σαΐντ. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τα πράγματα, κυρίως για τους επιβάτες, και να αποφύγουμε στη συνέχεια καταχρήσεις όσον αφορά τις εργασιακές ε, σχέσεις των εργαζομένων κυρίως. Δεν υπάρχει βεβαίως αμφιβολία ότι μια κάποια περαιτέρω απελευθέρωση μπορεί να είναι ένα στοιχείο το οποίο θα είναι προς όφελος αυτών των στόχων. Ε, σίγουρα όχι να είναι αυτοσκοπός η απελευθέρωση, αλλά να είναι το μέσο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτή τη διαδικασία και αυτή η διαδικασία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ελέγχεται. Ε, συμφωνώ λοιπόν με την παρέμβαση ε, του εκπροσώπου τη Επιτροπής των Περιφερειών για την ανάγκη να ενισχύσουμε τον Ευρωπαίο Ρυθμιστές ε, που είναι μία εκ των όνου κάνευ ε, προϋπόθεση προκειμένου να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο αντάξιο του ονόματός του και να μην έχουμε μόνο εθνικά συστήματα. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό και γιατί η απελευθέρωση δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Διότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με το θέμα των ε, κατασκευών ε, και τα κατάλληλα μέσα. Και δεν είναι απελευθέρωση σαν αυτή τη απελευθέρωση του φυσικού αερίου π.χ. Κατά την έποψή μου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση η οποία ε, όχι μόνο δεν στέκει αφεαυτής, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει και σε απόλυτο μονοπόλιο αν δεν προσέξουμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και να υπάρχει και κατάλληλο κόστος για τους επιβάτες. Ευχαριστώ, ο κύριος ε, Πανιό για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε απολύτω ότι ε, δεν είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί στις συζητήσει τις τελευταίες εβδομάδες και δεν το έχουμε λάβει δεόντω υπόψη. Έχουμε μια πολιτική συζήτηση η οποία θα έχει συνέπειες όχι μόνο για τους υπαλλήλους των σιδηροδρόμων αλλά και για όλους όσους εποφολούνται τη ε, πολιτική για του σιδηροδρόμους. Ακούω πολλέ φορέ και από ευρωβουλευτές ότι κυρίως θα πρέπει να θεωρούμε ότι έχουμε τεχνοκρατικά στοιχεία εδώ και θα πρέπει συχνά να στεκόμαστε σε αυτό. Και θα πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι ένα μοντέλο στο οποίο ο διαχειριστής των δικτύων και των υποδομών ανήκει σε ένα ενιαίο ε, όμιλος ε, ή μια ολοκληρωμένη υπηρεσία είναι πιο αποτελεσματικό. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη όμως που να αποδεικνύει ότι ο σαφής διαχωρισμός, ε, κύριε Πρόεδρε, όπως είπε και ο συνάδελφος Δομινί Κρικέ, θα είναι το καλύτερο μοντέλο από οικονομικής πλευράς, από πλευράς ανταγωνισμού του συστήματος και από πλευράς σιδηροδρόμων. Ε, το αντίθετο, από ό,τι φαίνεται, θα διαταρέξει την ε, σωστή λειτουργία και κυρίως σε κάποιες χώρες, θα πρέπει να υπενθυμίσω στις κάτω χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κάποιες νέες μορφές ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών των ε, δικτύων και των υποδομών χρησιμοποιούνται σε πειραματικό επίπεδο. Ε, θεωρώ ότι ο τελικός στόχος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των δικτύων και των υποδομών δεν συνάδει με τους οικονομικούς, κοινωνικούς στόχους μας και τις υπηρεσίες που θέλουμε να προτείνουμε το αύριο το πρωί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι αυτή η συζήτηση, είναι πολιτική η συζήτηση και αυτή είναι η ευκαιρία να την κάνουμε. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, και θεωρώ ότι οι τροπολογίες του συναδέλφου Σαϊντελ Κατράουι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση για να προστατεύσουν ε, και τους εργαζομένους στους υδροδρόμους αλλά και τους καταναλωτές. Ο κύριος Κάλιτσε και δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, ξέρω ότι πρέπει να ε, μιλήσω γρήγορα. Το είδα, Πρόεδρο, ότι με προσπεράσετε. Δεν πειράζει. Εδώ και δύο χρόνια προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις υδροδρομικές ε, μεταφορές. Πάντα κάτι βελτιώνουμε και πάντα κάτι υπάρχει για να βελτιωθεί ακόμη. Αν δούμε γενικώ τι σιδηροδρομικέ μεταφορέ και, και το διαχωρισμό μεταξύ των μεταφορών ατόμων και ε, αγαθών από, την, από τις υποδομές, θα δούμε ότι οι παρεχόμενες ε, υπηρεσίες ε, γίνονται χειρότερες αυτό δηλαδή που είχαμε κάνει καλά, ε, που θεωρήσαμε ότι το σχεδιάσαμε καλά, μετά από κάποια χρόνια είδαμε ότι δεν είχε τα σωστά αποτελέσματα. Το άνοιγμα της αγοράς είναι καλό, αλλά θα πρέπει να συνδεθεί με κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες. Σήμερα, στους σιδηροδρόμους της ε, Τσεχίας, εμείς δεν έχουμε δυνατότητες και έχουμε πολλές ε, σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και για τη μεταφορά ατόμων και για τη μεταφορά αγαθών. Αλλά οι δυνατότητες δεν υπάρχουν. Αν ε, θα πρέπει, αν πρέπει να συμπεριληφθεί κάποιο ε, άλλος, θα πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες των τσεχικών σιδηροδρόμων. Πώς θα γίνει αυτό με καλύτερη διαχείριση ίσως για τον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών. Σε είναι βέβαια αμφιλεγόμενο θέμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο το δίκτυο να διατηρηθεί. Έχουμε 13 περιφέρειες εμείς και κάθε περιφέρεια ζητάει κάτι διαφορετικό και στα όρια μεταξύ των διαφόρων περιφερειών ε, τελειώνει μια μεταφορά και αρχίζει επίσης μια μεταφορά. Και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα γιατί δεν μπορούμε να τα λύσουμε τα θέματα αυτά θεωρητικά. Πρέπει πρακτικά να παρέμβουμε. Για την έκθεση του κυρίου για τα σχόλιά σας, ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεση και για τις διάφορες τροπολογίες για την ε, οδηγία που δημιουργεί την, ε, τον ενιαίο συγκλονικό χώρο και την αναδιατύπωσή τη. Ε, όταν κάναμε τι διαπραγματεύσει, συμφωνήσαμε Συμβούλιο, Κομισιόν και Κοινοβούλιο ότι η αναδιατύπωση ήταν σημαντικό βήμα, αυτό που χρειαζόταν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την περαιτέρω εργασία για τη διακυβέρνηση. Και αυτό, περί αυτού ακριβώς πρόκειται στην πρότασή μας. Η πρότασή μας δεν μιλά για διαχωρισμό. Η πρόταση μιλάει για έναν πιο αποτελεσματικό ε, μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των ε, υποδομών. Αν δείτε για ένα, μια μπροσούρα που έχουμε ε, βγει και θα συζητηθεί σε 10 μέρες στο Ταλίν, δείχνει ότι ο διαχειριστής των υποδομών ε, δεν είναι προκύπτει μόνο από αυτή την πρόταση τη δική μα. Υπάρχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και σε εθνικό επίπεδο επίση υπάρχουν δραστηριότητε. Αλλά η ουσία τη πρόταση τη Κομισιόν είναι όντω να ενισχύσει το ρόλο του διαχειριστή υποδομών στην όλη ε, ανάπτυξη αυτού του συστήματο και την ολοκλήρωση του συστήματο των ε, σιδηροδρομικών μεταφορών. Αυτό ο διαχειριστή θα πρέπει να είναι ευρω... σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι το όλο νόημα και νομίζω ότι υποστηρίζεται από την Επιτροπή, βλέποντα και τι τροπολογίε. Βεβαίω ο διαχειριστή αυτό ε, και το, είπατε, το είπαν αρκετά ε, μέλη σα σήμερα, πρέπει να γνωρίζει τι ανάγκε των χρηστών του δικτύου των σιδηροδρόμων και επίση αυτό ο διαχειριστή θα είναι υπεύθυνο για όλε τι πτυχέ τη διαχείριση ε, υποδομών. Και ένα σημαντικό κομμάτι τη πρόταση τη Κομισιόν, που νομίζω ότι το υποστηρίζει και ο εισηγητή, είναι ότι έχουμε διευρύνει το, το πεδίο των λειτουργιών, των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή, έτσι ώστε να να, να μπορεί να παρέχει αποτελεσματικέ αποδοτικές υπηρεσίες και να μπορεί να ελέγχει και το κόστος που προκύπτει από όλε αυτές τις δραστηριότητε. Τρίτον, Βεβαίω ο διαχειριστή υποδομών είναι σημαντικό σημείο, το είπαν και αρκετοί ευρωβουλευτέ. Ο διαχειριστή λοιπόν αυτό πρέπει να είναι ανεξάρτητο, απολύτω πλήρω ανεξάρτητο, θα προσέθετα εγώ, και βεβαίω είναι πολύ πιο απλό αυτό να γίνει σε, μια, σε ένα αποσυνδεδεμένο σύστημα. Αλλά εμείς από τη δική μας την πλευρά δείχνουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό και εντός ενός ολοκληρωμένου συστήματος και διασυνδεδεμένου. Είναι κοινή λογική να δούμε και τις ε, ροές των ε, κονδυλίων, να αποφύγουμε να υπάρξουν ε, επιπλέον κονδύλια είτε δημόσια είτε άλλα προς, τους, προς τις ε, διαχειριστικές αρχές και βεβαίως αυτό θα το κάνουν οι ρυθμιστικές αρχές που επίσης ενισχύονται μέσω της αναδιατύπωσης. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο σήμερα να ρυθμιστούν αυτές οι ε, ροές κονδυλίων και γι' αυτό σήμερα προσπαθούμε να ενισχύσουμε ε, τις ρυθμιστικές αυτές αρχές και τον κλάδο. Οι διάφορες τώρα διατάξεις που αναφέρονται ως συνοικό τείχος επίσης είναι κοινή λογική για μας για να δούμε ποιος θα πάρει τελικά τις κλήρες αποφάσεις και θα εξασφαλίσει ότι όντως λειτουργούν τα πράγματα είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά και βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με θέματα ε, ε, μικτής ε, εμπορικής ενημέρωσης. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αρχή διαχειριστική των υποδομών μπορεί να λειτουργήσει και σε μια διασυνδεδεμένη δομή. Αλλά είναι σαφές ότι αν πολλές από τις τροπολογίες αυτές ε, που κυρίως, και κυρίως αυτές που θέλουν να διαγραφούν οι περισσότερες από τις διδάξεις που υπάρχουν στην πρόταση Κομισιόν διατηρηθούν, αυτό θα μας πάει πίσω. Θα μας πάει πίσω στην παλαιά ολοκληρωμένη δομή. Και ουσιαστικά αυτό θα σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις ε, ε, θα διαχειρίζονται σε έναν βαθμό τις υποδομές τους, θα μπορούν να αναπτύξουν, αλλά θα ήταν πολύ πιο, πολύ πιο δύσκολο να πούμε ότι οι, α, ε, ε, υποδομές βελτιώνονται για το καλό όσων τις χρησιμοποιούν. Μετά, ε, για το άνοιγμα της αγοράς. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της πρόσβασης στην αγορά και των υποχρεώσεων προς τους πολίτες, παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η συνάδελφό μου θα ε, σχολιάσει το θέμα αυτό, αλλά αν δείτε τη διασύνδεση μεταξύ των δύο, νομίζω ότι η ισορροπία έχει να κάνει με το πώ θα ενισχύσουμε τον, ε, τον ε, ανταγωνισμό για, την, για, τον, για τους υδροδρόμους που αποτελούν μονοπόλιο για πολλά κράτη χώρα, πώς κρατεί μέλη, πώ θα ενισχύσουμε την καινοτομία, πώς θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, πώς θα ενισχύσουμε τους χρήστες των σιδηροδρόμων και η ισορροπία βρίσκεται μεταξύ των δύο ε, εκθέσεων ουσιαστικά. Δηλαδή, η, ε, τι γίνεται με τους διαγωνισμούς για τις ε, υπηρεσίες που πρέπει να διατηρηθούν και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την πρόσβαση στην αγορά. Αν περιορίσουμε την πρόσβαση στην αγορά, αυτό θα πρέπει να γίνει με το μικρότερο δυνατό κόστος. Βεβαίω θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει και το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά αυτέ τι τροπολογίε για τι ε, δημόσιε υπηρεσίε στου σιδηροδρόμου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριο Γκρό. Αν θέλουν οι συγκητέ θα πάρουν ε, το λόγο στο τέλο. Πάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Γκρό για τον κανονισμό για το άνοιγμα τη αγορά εγχώρων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μας ε, η προϋπόθεση, η βασική, είναι ότι με αυτή την πρόταση ε, θέλουμε να βελτιώσουμε τι ε, δεν λειτουργεί, αλλά όχι να καταστρέψουμε αυτά που ήδη λειτουργούν. Για την αποδοτικότητα τώρα ε, μιλούμε για τα κράτη-μέλη, για τις περιφέρειες οι οποίες θα πρέπει να συμβάλλουν οικονομικά και ο ανταγωνισμός για μένα έχει αξία μόνο στο βαθμό που τα δημόσια κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο και να μην δημιουργούνται σχέσεις κάτω από το τραπέζι. Ε, θα θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τις ε, τροπολογίες τους, 382 συγκεκριμένα μου υπέβαλαν, πολύ καλές οι προτάσεις, να πω ότι θεωρώ ότι τις, μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες προτάσεις, γι' αυτό για τις ε, τροπολογίες που προτείνουν διαγραφή δεν μπορώ να συμφωνήσω, θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Τώρα κάποια σημεία συζητήθηκαν ήδη, ο ορισμός ε, για την δημόσια αρχή, τα ακούσαμε ήδη από την Επιτροπή των Περιφερειών και... Ε, και εγώ είμαι υπέρ των ε, διασυνοριακών της διασυνορικής πτυχής. θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο ορισμό ώστε αυτό που μπορεί να λειτουργήσει να μην γίνεται αδύνατο να λειτουργήσει. Το πεδίο εφαρμογή τώρα για, και, οι κοινό, και ε, κοινέ ε, υποχρεώσεις, ε, οι τροπολογίες που μιλούν για την απόδοση, για την αποδοτικότητα συγγνώμη, των δικτύων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Τώρα, υπάρχουν κάποιες ε, πτυχές για τις ε, διασυνοριακές ε, μεταφορές, τις είπαν οι συνάδελφοι, η διατροπικότητα, οι αρμόδιες αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, να μην δημιουργήσουμε εδώ πέρα σύγκρουση συμφερόντων. Πρέπει βεβαίω όσοι συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο και συμμετέχουν να μπορούν να έχουν λόγο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ανώτατο όριο και το εύρο των δημοσίων υπηρεσιών και των σχετικών συμβάσεων, θα πρέπει εδώ να έχουμε σωστή ισορροπία μεταξύ μικρών και μεγάλων κρατών. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα να φτιάξουμε μία ενιαία διάταξη. Μια χώρα όπως η ε, Γαλλία ή το Λουξεμβούργο δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο ίδιο πλαίσιο. Ε, τώρα για τις κοινωνικές ρυθμίσεις ε, είχα, έλαβα κάποιες ε, τροπολογίες. Ε, υπήρξε και η σχετική ε, συμφωνία με την ETF που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Για την αμοιβαιότητα τώρα, εγώ είμαι υπέρ της αμοιβαιότητας. Θα πρέπει να γίνεται από τις χώρες όμως η αμοιβαιότητα αυτή. Θα πρέπει να είναι δυνατόν τα, οι συμβάσεις που δίνονται να μην καταλήγουν σε μονοπόλια. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ε, συζήτηση που πρέπει να κάνουμε εδώ. Τώρα για τις τρίτες χώρες ε, θεωρώ ότι πρέπει να είναι δυνατόν, αλλά δεν, μπορούν να, δεν μπορούμε να τις υποχρεώσουμε. Άμεσες τώρα συμβάσεις, αυτό είναι ένα θέμα γενικό. Άρθρο 5 παράγραφος 6 έχει διαγραφεί και έχουν προβλεφθεί κάποια άλλα πράγματα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο τρόπος ε, ε, απόδοσης των συμβάσεων θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και πρέπει να δούμε αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος ή αυτή. Αν, κάποιος, ε, αν κάποια διαδικασία έχει καλά αποτελέσματα και το έχουμε δει και στο παρελθόν, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι μιλούμε πάντα με, για διαφανείς ε, τρόπους και κυρίως ό,τι αφορά τις άμεσες, ε, ε, τους, τους διαγωνισμούς με, άμεση με άμεσο ανάδοχο. μιλούμε για πάρα πολλά εκατομμύρια κονδύλια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Και κλείνοντας πρόεδρε να πω ότι οι, δια, που αφορούν την μεταβατική περίοδο είναι σημαντικές γιατί μιλούμε για ένα σύστημα μέχρι το 2029. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τι εμπειρίε που έχουν κάποιε χώρε και κάποιε όχι. Αύριο θα, ε, ε, την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η πρώτη συνάντηση με του σκιώδει. Ε, ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση. Ελπίζω ότι τήρησα το χρονοδιάγραμμα που μου βάλετε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Ισηγητά, συνάδελφοι. Θα μιλήσω και εκ μέρου ε, του κυρίου Λιμπεράτσκι που είναι ο σκιώδη μας. Ευχαριστεί τον ε, συνάδελφο για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Ήταν πολύ επικοδομητική συνεργασία που έχει υπάρξει μέχρι στιγμή. Ο κύριος Λιμπεράτσκι ε, σημειώνει ότι πριν από τέσσερι ημέρε η πολωνική μετάφραση των τροπολογιών έφτασε στα χέρια του ε, και επομένως ε, δεν μπορούσε να διαβάσει αυτές τις 238 ε, σελίδες τροπολογιών, γι' αυτό ζητά συγγνώμη. Πραγματικά είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους οι τροπολογίες. Πολλές μιλούν για διαγραφή, για τα κατόφλια κτλ. Για κάποιες τροπολογίες τα κατόφλια για, τις ε, άμεσες, ε, για τους άμεσους αναδόχους έχουν αυξηθεί. Οι, αυτές οι δυνατότητες θα πρέπει να υπάρχουν μόνο σε ε, πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, γι' αυτό δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει λόγος να υπάρξει αναθεώρηση στα πλαίσια της εφαρμογής της 13-17. Αυτό βεβαίως δεν έχει να κάνει με τον ρόλο που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να έχει ένας δημόσιος φορέας. Τώρα, η ε, Επιτροπή είναι υπέρ της αναθεώρησης ε, για τα, για τα PSOs. Ε, θα πρέπει να δούμε όμως, μέχρι τις 26 Νοέμβρη μπορούμε να τα καταφέρουμε, να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό. Και επίσης, ο πυρήνας της πρότασης της Κομισιόν θα παραμείνει ανέπαφος και αν τελικά πάει στην Ολομέλεια η αναδιατύπωση και αν η Κομισιόν συνεχίσει την πρότασή της, ίσως να πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις μονοπωλιακές αγορές. Ο πυρήνας της πρότασης Κομισιόν πέραν της ε, απελευθέρωσης ε, των αστυνομικών ε, μεταφορών έχει να κάνει και με την κοινωνική διάσταση αυτού του κανονισμού. Γιατί αν δεν τα καταφέρουμε η 1370 του, 7, του 2007 να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων κτλ. τότε δεν ξέρω, μπορώ ίσως να χρειαστεί να στείλουμε πίσω την πρόταση της Κομισιόν στο σύνολό της. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν στα βασικά, στα ουσιώδη της ε, υπόθεσης και αυτά είναι τα τεχνικά κομμάτια που αφορούν στο τέταρτο πακέτο. Ευχαριστώ. για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Γκρό, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ τον εισηγητή και για το έργο του και για την αγαστή συνεργασία και προσβλέπω στι συνεδρίε που θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι ο στόχο είναι κοινό, να βελτιώσουμε την ποιότητα τη δημόσια υπηρεσία προ του πολίτε μα, διότι όλοι λαμβάνουμε διαμαρτυρίε από του πολίτε για την κατάσταση των σιδηροδρόμων, για το πώ είναι πάντα καθυστερημένα τα, τρεάν, τα τρένα, δεν είναι καθαρά και το πώ επιδεινώνεται η, περιοχή, η ποιότητα των υπηρεσιών κάθε χρόνο. Πρέπει να δράσουμε λοιπόν πλέον. Είναι η σειρά μας να ανοίξουμε πλέον την αγορά το συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό ακριβώς εμείς οι φιλελεύθεροι είμαστε ε, ευχαριστημένοι με την ημερομηνία που προτείνει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Προτείνουμε την ε, προθεσμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2019 και θεωρούμε ότι η προθεσμία για το 2029 για την υποχρεωτική ε, δυνατότητα προκήρυξης διαγωνισμών χωρίς άμεση ανάθεση είναι ε, πολύ με καθυστερημένη. Όσον αφορά τώρα τους ε, διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί κατά την άποψή μας θα πρέπει να γίνεται απευθείας ο κανόνες και η άμεση ανάθεση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε να περιοριστεί η διάρκεια των συμβάσεων που ανατίθεται με άμεση ανάθεση. Να σας υπενθυμίσω την τροπολογία 19 των συναδέλφων Ντεμπάκερ και Μπένιν που ζητούν ε, ένα όριο 5 ετών. Κατά τη μεταβατική περίοδο, η οποία ελπίζουμε ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη φυσικά, θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή και τους συναδέλφους να δουν την τροπολογία μου 339 για να μπορέσουμε να δώσουμε και ρόλο στη ρυθμιστική αρχή. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αιτιολογούν την επιλογή σε περίπτωση άμεσης ανάθεσης και θα αποστείλονται και σχετικές αιτιολογίες στον ρυθμιστή, στον ανεξάρτητο ρυθμιστή για να δίνει την έγκρισή του. Τώρα από εκεί και πέρα τη δυνατότητα ε, της... Ε, ε, ικανοποίηση των πελατών θα πρέπει να είναι βασικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη κατά την άμεση ανάθεση. Επίσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποτελέσουμε προτεραιότητα για να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού ε, στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να δεχτείτε κάποιες από αυτές τις ιδέες στο συμβιβασμό. Ευχαριστούμε κύριε Τρεμόσα. Ο κύριος ε, Ζαρίμπη, εκ ονόματος των Πρασίνων, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Ματία Γκρός, τον εισηγητή μας, για το πνεύμα ε, συνεργασία το οποίο έχει επιδείξει και για τα όσα έχει κάνει σε αυτό το τόσο περίπλοκο και από τεχνικής αλλά και από πολιτική σκοπιά ζήτημα. Είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ε, κάποιοι αναφέρονται και στι διάφορε ευαισθησίε. Θέλουμε να βελτιώσουμε την προσφορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα χωρί να διακυβεύεται η ασφάλεια η οποία μα ενδιαφέρει όλου για τα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά συστήματα και θέλουμε να λάβουμε υπόψη και τι κοινωνικέ συνθήκε. Νομίζω ότι αυτή είναι η έννοια και κάποιων τροπολογιών που ε, κατατέθησαν προς αυτά τα θέματα και ε, κυρίως θέλουμε να υπάρχει και συλλογικό πνεύμα και ευαισθησία. Ε, να πω κύριε Πρόεδρε ότι θεωρώ ότι υπάρχει κάποια πρόοδος ε, και χαίρομαι γι' αυτό. Κυρίως ε, το θέμα των κοινωνικών στοιχείων που είναι πολύ σημαντικό διότι μας ενδιαφέρει το θέμα των υπαλλήλων και το αν θα προσλαμβάνονται όταν η, αγορά θα περνάει από τα χέρια του ενός παρόχου σιδηροδρομικών υπηρεσιών στον άλλον. Θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται και να λαμβάνεται υπόψη και επικουρικότητα και συλλογικές συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο για σιδηροδρομικούς υπαλλήλων, για να γίνονται επίση και σεβαστά και κάποια κοινωνικά πρότυπα, τα οποία θεωρώ ότι είναι θεμελιώδη. Υπάρχει και μια κάποια πρόοδος, κατά την άποψή μου, για τον ορισμό της αρμόδιας τοπικής αρχής, η οποία είχε ληφθεί υπόψη στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση να επιστρέψουμε στον αρχικό ορισμό. Ε, θέλουμε να έχουμε ένα πάροχο σε τοπικό επίπεδο λοιπόν, κάποιον ο οποίος θα διαχειρίζεται τις μεταφορές ε, τις σιδηροδρομικές εκεί. Και επίσης ε, υπάρχει και μια αύξηση του επίπεδου εδώ και από την πρόταση του ίδιου του εισηγητή και από τις διάφορες τροπολογίες που κατατέθησαν, διότι έτσι φαίνεται ότι θέλουμε να έχουμε ε, μια στρατηγική εικόνα της λειτουργίας σε τοπικό επίπεδο. Και υπάρχει και ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι αποτελεί φραγμό, το θέμα της αμεβαιότητας, το οποίο δεν έχουμε ακόμα διαχειριστεί επαρκώς, πρέπει να το τελειοποιήσουμε και να αντιληφθούμε καλύτερα την έννοια. Για τις τρίτες χώρες δεν υπάρχει πρόβλημα. Αμοιβαιότητα μεταξύ χωρών ε, είμαι αντίθετος. Για αμοιβαιότητα μεταξύ ε, αρχών είμαι υπέρ. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα δεν είναι δυνατόν να απαγορεύσουμε σε κάποιον να δραστηριοποιηθεί σε μια αγορά σε διάφορες ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η προθεσμία που ε, προτείνεται το 2029, κάποιοι λένε ότι είναι πολύ καθυστερημένη. Θα χρειαζόμαστε όμως και χρόνο να προσερμιστούμε. Εγώ είμαι υπέρ. Ε, θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε και μια ενδιάμεση λύση μεταξύ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πρότασης του εισηγητή. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσω εδώ και να σας υπενθυμίσω και την τροπολογία μου 315 για την άμεση ανάθεση, όπου προτείνω και μία εναλλακτική λύση, να λαμβάνετε υπόψη και η τεχνική και η οικονομική προσφορά για να μπορεί ένας αρμόδιος τοπικός φορέας να αναλάβει απευθείας ε, τη διαχείριση ενός δικτύου. Ο κύριος Ζήλε για τρία λεπτά. Τσέλερ, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ματιό Γκρός. Εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο και με ιδιαίτερα οργανωμένο τρόπο που μας παρουσιάζει τώρα τα πορίσματα της εργασίας Το Ελπίζω μετά τις συζητήσεις να καταλήξουμε και σε μια συμβαστική λύση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είναι αλληλένδετες αυτές οι δύο εκθέσεις που μας έχουν απασχολήσει μέχρι στιγμής, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να προσέξουμε όταν ανοίγουμε τις, και απελευθερώνουμε τις αγορές ε, θα πρέπει να διατηρούμε ε, τα συστήματα απόδοσης ε, ευθυνών για τους φορείς παροχής δημοσίων υπηρεσιών καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών. Εσείς αναφερθήκατε στις διαφορές ανάμεσα στη Γαλλία και το Λουξεμβούργο. Ναι, αληθεύει αυτό, αλλά όπως αληθεύει και για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιώκοντας ε, την ε, ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών δικτυών θα πρέπει όντως να λάβουμε υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Για τη μεταβατική περίοδο θα συμφωνήσω με τους φιλελεύθερους ε, το να ορίσουμε την ημερομηνία το 2029 δείχνει έλλειψη σοβαρότητας κατά τη δική μας άποψη. Θα θέλουμε να περιοριστούμε το 2019 αυτό που είχε προτείνει αρχικά εξάλλου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το θέμα της αμοιβαιότητας έχω κάποιους συνδυασμούς, κυρίως όταν ε, λαμβάνω υπόψη αυτό που μας λένε οι εμπειρογνώμονες ε, στον τομέα αυτό. Εάν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσουμε να αποκλείσουμε κάποιους φορείς και ταυτόχρονα δεν επιτρέπουμε σε μεγάλους ιδιωτικούς φορείς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισέλθουν ε, στην αγορά τρίτων χωρών. Ε, έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να μην πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι στην ομοθέσια που θεσπίζουμε. Αν πραγματικά επιδιώκουμε μια δέσμη ομοιόμορφων νομοθετικών μέτρων δεν θα πρέπει Ε, να διαλέξουμε δρόμο διαφορετικό από το, την κοινή προσέγγιση ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αναγνώριση των νομοθετικών μας διατάξεων. Οι φιλελεύθεροι έχουν υιοθετήσει λοιπόν αυτή την στάση. Εάν δεν προστατεύσουμε ε, την αγορά μας και αν δεν ζητήσουμε ρήτρε αμοιβαιότητας από τις τρίτες χώρες, τότε όντως θα υποστούμε απώλειες. Δύο είναι τα τεινά με αυτή τη ρήτρα αμοιβαιότητας. Ε, οι σχέσεις στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Δύο διαφορετικά πράγματα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ρωτήσω τον κύριο Κράμερ ε, ποιος θα ε, θέλει να πάρει τον ελάχιστο μισθό για να δουλεύει και βάρδιες ε, κύριε Κράμερ. Χρειαζόμαστε κοινωνικά πρότυπα στον κλάδο των σιδηροδρόμων. Σχόλια του κύριου Κράμερ εκτός ε, μικροφώνου. Λοιπόν, η δική μου ομάδα για την ε, τροποποίηση για τους ε, PSOs είναι αντίθετη. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί βεβαίω η συζήτηση και τα κράτη-μέλη πρέπει από το 2014 στο 2015 να υποβάλουν μια ενδιάμεση έκθεση. Η τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας ακόμα τρέχει, οπότε θεωρούμε ότι η αλλαγή του κανονισμού είναι πάρα πολύ νωρί για να γίνει τώρα. Ε, έχουμε υποβάλει υπό ε, τροπολογία για ε, να πάει πίσω η πρόταση της Κομισιόν. Από την ECR και από τους σοσιαλιστές επίσης έχουν συνυπογράψει οι συνάδελφοι. Βεβαίως έχουμε υποβάλει και άλλες τροπολογίες για να συμμετέχουμε και επί τη ουσία τη συζήτηση. Σημαντικό είναι εδώ το εξή. Η εγγυημένη αρχή μέσω του πρωτοκόλλου 26 της Συνθήκης Λισαβόνας ε, για την αριθμιστική ε, αρχή σε ό,τι αφορά τις ε, διάφορες δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να διτηρηθεί. Τώρα, για τις διάφορες επιχειρήσεις και το πεδίο λιγμών που έχουν, αυτό λέει η πρόταση ότι θα μειωθεί. Πρέπει να υπάρχει σωστή απόδοση, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες, αποδοτικές και δεν πρέπει να τις διακυβεύσουμε σε έναν διαγωνισμό προφανώς θα ε, επιλεγεί ο πιο φτηνός και όχι ο καλύτερος. Και αυτό βεβαίως θα, υπάρξει, θα σημαίνει κόστος σε περισσότερο για τους ε, πελάτες των σιδηροδρόμων. Οπότε η αρχική εκδοχή του άρθρου 5.6 του κανονισμού 1370 του 2007 θα πρέπει να παραμείνει ως έχει γιατί προσφέρει στα κρατημέλη την απαραίτητη ευελιξία και ευτυχώ το βλέπουν και, άλλες, ε, και άλλοι ε, συνάδελφοι από άλλε ομάδε ε, με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να έχουμε ποιοτικέ υπηρεσίε. Τα κοινωνικά πρότυπα επίση παίζουν σημαντικό ρόλο για μα και γι' αυτό έχουμε υποβάλει τι σχετικέ τροπολογίε. Είμαστε επιπισμένοι ότι η κοινωνική προστασία αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών στους σιδηροδρόμους και οι δεσμευτικές, ε, προϋποθε... οι διατάξεις ε, και για την άμεση ανάθεση αλλά και για τους διαγωνισμούς θα πρέπει να ισχύουν. Η κοινωνική προστασία θα πρέπει να ε, υπάρχει είτε μέσω του εθνικού, της εθνικής νομοθεσίας είτε μέσω των τομεακών δασμών και επίσης θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική μεταφορά προσωπικού έτσι ώστε να υπάρχει επαρκές προσωπικό για να μπορούν να παράγονται αυτές οι υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Έχω ακόμα έξι ομιλητές. Επτά με τον κύριο Κόλιτσεκ. Και κλείνουμε αυτό τον κατάλογο γιατί αλλιώς... Ξέρω μιλάτε εκ μέρους του κύριου Λιμπεράσκη, αλλά βοηθήστε με αν θέλετε. Okay, for minutes each. Για δύο λεπτά ο καθένας, ε, για να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Ελκαντράου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Γκρός. Νομίζω ότι θα συνεργαστούμε αρκετό καιρό, διότι υπάρχει σαφής ε, σχέση μεταξύ της έκθεσής του και της δικής μου. Τώρα θα ήθελα να περιοριστώ και να πω δύο λόγια για τις τροπολογίες που κατέθεσα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το κείμενο να αναφέρεται και στην κοινωνική πτυχή. Να ενισχύσουμε μάλιστα αυτή την πτυχή. Παραδείγματο χάρη, κατά τον σχεδιασμό των μεταφερικών σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ε, η κοινωνική προστασία και οι συλλογικές συμβάσεις ε, οι οποίες είναι ενισχύ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Όποιος θέλει να παρέχει αντίστοιχε ε, υπηρεσίες βάσει συμβάσεων δημοσίων ε, υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις συλλογικέ συμβάσει. η διαφορά μεταξύ της άμεσης ανάθεσης και της προκήρυξης διαγωνισμών. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη ευελιξία και να σκεφτούμε λίγο καλύτερα το σχεδιασμό μας, ιδίω για μεσαίου μεγέθους χώρες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και πώς έχει η πραγματική κατάσταση επιτόπου. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε και τι γίνεται σε χώρες μεταξύ, ε, που έχουν μεταξύ 10 και 15 χιλιάδε τετραγωνικά χιλιόμετρα θα πρέπει να υπάρχει, μπορεί να υπάρχει ένας πάροχος και να υπάρχει δυνατότητα έμεση ανάθεσης ή να λαμβάνουμε υπόψη τον όγκο των επιβατών που επεξυπηρετεί κάποιος. Θα πρέπει έτσι να μπορέσουμε να έχουμε ένα ισχυρότερο δίκτυο και έτσι θα καλύπτεται και μεγαλύτερη απόσταση. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες πτυχές. Θα τα αφήσω σε αυτό το σημείο προς το παρόν. Ε, θέλουμε να εξετάσουμε και το θέμα της αμοιβαιότητας και της άμεσης ανάθεσης, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε αυτό. Ο κύριος Ρικέ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρός. Είναι αξιοσημείωτη δουλειά του, είναι και ο Ε, είδα και την έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία τονίζει ένα βασικό στοιχείο στο θέμα των μεταφορών θα μπορέσουμε να βρούμε την ισορροπία στα συγκεκριμένα μέτρα, διότι θα μπορέσουμε να καθορίσουμε επακριβώς και τους στόχους ε, των μεταφορών και όπως είπε προηγουμένως και ο Σαΐδ, να έχουμε και κατάλληλους κανόνες για κοινωνική προστασία και για το προστασία του περιβάλλοντος και να έχουμε και ένα σχέδιο μεταφορών. Αυτό θεωρώ είναι πολύ σημαντικό για όλες μας τις ε, ε, διατάξεις νομοθετικές. Όσον αφορά τώρα τον όγκο των υπηρεσιών για τις βάσεις ε, παροχής δημοσίων υπηρεσιών και την άμεση ανάθεση, είναι διαφορετική η κατάσταση σαφώς, είναι διαφορετικό το Λουξεμβούργο και διαφορετική η Γερμανία και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ένα περιφερειακό ε, κατόφλι και όχι εθνικό κατόφλι. Ε, νομίζω ότι είναι μια καλή κλίμακα διότι έτσι θα έχουμε και το μεγάλο πλεονέκτημα να μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλύτερα ε, εξέταση επιτόπου είναι καλή ευκαιρία, θα είναι μια χαμένη ευκαιρία διότι δυσκολευόμαστε να βρούμε τις κατάλληλες ισορροπίες, θα πρέπει να βρεθούμε ε, ε αντιμέτωποι και με τις εθνικές δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν. Όσον αφορά τις ε, προθεσμίες, να πω στον εισηγητή νομίζω ότι το 2029 είναι πολύ μακριά, θα πρέπει να βρούμε κάτι ενδιάμεσο, θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του 2019 και του 2029, αλλά το 2029 είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και ένα τελευταίο όσον αφορά την κοινωτική αμοιβαιότητα. συνάδει αυτό με την συνθήκη και με το πνεύμα των συνθήκων και με όλες τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Κατά την άποψή μου θα υπάρξει ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να προβλέψει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν τη σοφία της. Νομίζω ότι δεν έχει ακόμα επιλυθεί διότι υπάρχει θέμα εδώ πέρα ασυνέπειας. Ο κύριος Καντσιά για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρός. Πολύ συγκεκριμένα θα ήθελα να σταθώ σε πέντε σημεία για τα οποία έχω υποβάλει και τροπολογίες. Το πρώτο είναι το σημείο που αφορά την οικονομική ισορροπία, την οποία θα πρέπει να βρούμε μεταξύ του ανοίγματο τη αγορά και ε, των ε, διαχειριστών των συστημάτων. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο είναι το θέμα τη εσωτερική και εξωτερική αμοιβαιότητα, οι οποίε θα πρέπει να ρυθμίζονται από το κράτο μέλο, διότι υπάρχουν διάφορε καταστάσει στα κράτη-μέλη και κατά την άποψή μου για μένα αυτό θα ήταν υποχρεωτική φύσεω, διότι αλλιώ δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα την υποχρέωση προκήρυξης διαγωνισμός. Εγώ είμαι υπέρ ε, της προκήρυξης διαγωνισμών για την ανάθεση των συμβάσεων και ε, ένα τελευταίο σημείο είναι οι ημερομηνίε. Έχουμε τα κατόφλια, έχουμε τις καταληκτικές ημερομηνίε και θα πρέπει όλα αυτά ε, να μην τα θέσουμε σε αβέβαιες και πολύ μακρές διαδικασίες, διότι ουσιαστικά ελοχεύει ο κίνδυνος να παραβιάσουμε τις αρχές τις οποίες Τέλος, ο τεχνικός πυλώνας. Εγώ είμαι πέρα της απλούστευσης και της κεντρικής ε, ε, δυνατότητας ε, και για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων και για την έγκριση των ε, σιδηροδρομικών οχημάτων ε, και να έχουμε εκεί μεγαλύτερη ισχύ γιατί έτσι θα έχουμε και έναν Ευρωπαίο ρυθμιστή ο οποίος θα είναι πιο ισχυρός. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Γκρός για τη δουλειά που έχετε κάνει. Εξακολουθώ εγώ να ανησυχώ για τις τροπολογίες που προτείνουν το 2029 ως καταληκτική ημερομηνία. Ξέρουμε ότι αυτό το σε εφαλτήριο θα είναι και ότι θα χρειαστούμε χρόνο στην επόμενη γενιά μέχρι που να πλησιάσουμε καν την ολοκλήρωση της αγοράς. Οπότε ας στοχεύσουμε καλύτερα το 2019 για να αρχίσει η διαδικασία για το ανώτατο μέγεθος ε, για την υποχρέωση παροχή δημόσιας υπηρεσία. Ο κ. Δεμπάκη και ο υποφαινόμενο καταθέσαμε μια καταφαινόμενα πολυσύνθετη τροπολογία, αλλά η οποία όμω ακολουθεί το πνεύμα της τροπολογία του κ. Χαντρέου για το bundling. Θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτή τη λύση η πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το ζήτημα, αν μου επιτραπεί να, ερμηνεύσω το πνεύμα αυτής της πρότασης, μπορεί να οδηγήσει κάποια κράτη-μέλη να αισθανθούν ότι ε, τα όρια ε, προσδιορίζονται ακριβώς ε, από πάνω ή κάτω των εθνικών ορίων. Ίσως αυτό να αποτελέσει λύση. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσουμε για συγκεκριμένα όρια, θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε και ενδεχομένω να καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει. Για το ζήτημα τώρα των δημοσίων διαγωνισμών ε, κατά τη διαστολή με την ε, άμεση ανάθεση, θα έλεγα ότι οι διαγωνισμοί μας προσφέρουν ε, προσφέρουν όλες τις εθνικές αρμόδιες αρχές ευελιξία. Βεβαίως, Κύλουν οι διαγωνισμοί ως προς τη διάρθρωση και το μέγεθός τους. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανησυχούμε και να ακολουθήσουμε πλήρως αυτή την οδό των διαγωνισμών. Ε, θα έπρεπε να περιορίσουμε τη χρήση αυτού του μέσου ως προς το πεδίο εφαρμογής και τα όρια που θα θέσουμε. Ε, και συμφωνώ με τον κύριο Τσέλερ για τα όσα μας είπε για την αμοιβαιότητα. Ευχαριστούμε. δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Μάτιο Εγκρό. Άρχισε την παρέμβασή του λέγοντα ότι δεν πρέπει κανεί να χαλάει αυτό που λειτουργεί, οπότε ε, νομίζω ότι έτσι αναιρούνται οι τροπολογίε που κατέθεσαν από του σκιώδες. Εγώ θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να καταστήσουμε πνευματικότερου του Ευρωπαϊκού σιδηροδρόμους με αυτόν τον τρόπο, αλλά με τη συστηματικοποίηση ε, των λύσεων και με την μη διαβούλευση για τα επιμέρου όρια πορεία κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε μια χαοτική κατάσταση επιτόπου είτε ε, στα δίκτυα που χρησιμοποιούνται, τα, τα πυκνότερα δίκτυα και αυτά που ε, χρησιμοποιούνται πιο πυκνά σε κάποια κράτη-μέλη ή για συγκεκριμένα δρομολόγια. Ε, κινδυνεύουμε να γίνει ένα big bang ας πούμε και ταυτόχρονα να μην αυξηθεί η ζήτηση εμείς αντιπροτείνουμε τον ανταγωνισμό να τον επιδιώξουμε ως προς την διαχείριση, ούτως ώστε να υπάρχουν ανταγωνιστικές συμβάσεις διαχείρισης που θα υπάγονται στους όρους παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να καταγερματίζουμε τις επιχειρήσεις σε μικρά κομμάτια ή να αντικατασταθεί στο πέρας της σύμβασης η επιχείρηση. Μόνο η κεφαλή, η διοίκηση πρέπει να αντικατασταθεί, το πελώριο πλεονέκτημα Τη τη είναι να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη λειτουργία των πυκνότερων συχνά δικτύων. Ευχαριστούμε. Κράβαρ δύο λεπτά. Καταρχά να πω ότι είναι απαράδεικτο όταν μιλούμε για πάνω από 300 ή 200 ε, τροπολογίες θα τις παίρνουμε στην ε, γλώσσα μας ε, τρεις μέρες πριν τις συζητήσουμε. Οπότε, Πρόεδρε, προσπαθήστε με κάποιο τρόπο να έχουμε τις τροπολογίες τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν στη γλώσσα μας γιατί τελείως δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Είμαστε και εμείς πιεσμένοι. Ξέρουμε και η Κομισιόν και το Συμβούλιο παίρνουν το χρόνο τους για να διαβουλευτούν. Για αυτούς δεν έχει πολύ νόημα ο χρόνος ή ο μήνας, αλλά εμάς μας πιέζουν. Έχουμε λοιπόν ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο λέμε ότι θα λύσουμε το ε, ναι, ή, θα, δεν έχουμε πρόβλημα, ή έχουμε πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Δεν γίνεται να έχουμε ένα πρόβλημα και περιμένουμε το 29. Παρατηρείτε λοιπόν ότι ε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα, αλλά για μένα το σημαντικό είναι η αμοιβαιότητα στις ε, αναθέσεις. Ε, Υπάρχει μια αρχή. Βεβαίω ε, δεν θεωρώ ότι οι ιαπωνικέ εταιρείε μπορούν να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά όταν εμεί δεν μπορούμε να μπούμε στη δική του. Αλλά πάλι δεν συμφωνώ με το ότι η RTP ε, να παίρνει μια άμεση ανάθεση μια άμεση ε, στη χώρα τη μια άμεση σύμβαση και μετά να μπορεί να πάρει μέρο σε ένα διαγωνισμό για να αναλάβει το, το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τις ε, άμεσες αναθέσεις. Παίρνουν άμεσες αναθέσεις ακόμα και στη Γερμανία, που μάλιστα επιδοτούνται και κρατικά, και μετά μπορούν να κάνουν και προσφορές πιο φτηνές σε άλλες, σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό είναι πραγματικά διακριτική μεταχείριση, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει αυστηρή ε, αμοιβαιότητα για τις εταιρείες, για τις θηγατρικές εταιρείες. Φυσικά θέλουμε ε, ανταγωνισμό, πρέπει να υπάρχουν ελάχιστοι μισθοί, θέλουμε να προσφέρουμε ό,τι είναι καλύτερο, εγώ πολλές φορές ε, λέω ότι δεν έχω τόσα λεφτά και προφανώς ε, πρέπει να κάνω οικονομία. Ε, το, το πιο φτηνό είναι καλύτερο. μπορεί πολλές φορές η καλή ποιότητα να μην είναι τόσο καλή όσο να επιτύχει κανείς μια φτηνή τιμή. Αυτά από μένα. Ο κύριος Κόλιτσεκ για δύο λεπτά. E, ta neférová konkurence, o které se tady kolega zmiňoval, tu už máme. Ναι, για τον θέμητο ανταγωνισμό που είπε και ο συνάδελφος, υπάρχει και στην Τσεχία τέτοια κρούσματα. Οι μεγάλοι αγοράζουν σιγά σιγά τους μικρούς. Λοιπόν, τώρα επί της ουσίας. Η ουσία αυτής της έκθεσης ουσιαστικά βρίσκεται στην διασφάλιση των κοινωνικών προτύπων και στην διατήρηση της κυκλοφορίας ως δημόσιο αγαθού. Ε, τα όρια, ναι, πρέπει να οριστούν ανάλογα με το μέγεθος ε, της χώρας, ε, όπως, είπε και, όπως λέει και ο εισηγητής. Όχι από 10 εκατομμύρια χιλιόμετρα, αλλά από 35 εκατομμύρια. Στην περιφερειακή ε, στις περιφερειακές ε, μεταφορές οι ιδιωτικές εταιρείες ε, θέλουν να μπορούν να επιλέγουν. Δηλαδή οι περιφέρειες προσφέρουν ένα πακέτο, όχι μόνο ε, ένα δρομολόγιο, αλλά ένα ολόκληρο πακέτο, ένα κομμάτι του δικτύου των των, μεταφορών και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται και η λύση γιατί είναι κάτι πρακτικό που το βλέπουμε και καθημερινά να εφαρμόζεται, δεν είναι μια θεωρία. Ο πελάτης λοιπόν βεβαίως πρέπει να μπορεί να λάβει καλύτερες υπηρεσίες για την αμοιβαιότητα τώρα. Ε, μεταξύ ημών και της ε, Πολωνίας λειτουργεί αμοιβαιότητα και εδώ δεν προσπαθούμε να υποχρεώσουμε κάποιον να, είναι να δείξει αμοιβαιότητα απέναντί μας. Ε, οι πιο, οι πιο σύντομες ε, προθεσμίες μπορεί να βρίσκονται ε, σε αντίθεση με το όσα προβλέπει ο κανονισμός. Ίσως καλό θα ήταν να έχουμε μια ενδιάμεση έκθεση για το 2015 και μετά να προσαρμόσουμε τις ε, προθεσμίες. Είναι καλύτερο να έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη προθεσμία ε, από το να έχουμε μια πιο σύντομη για να, και να μην μπορούμε να την τηρήσουμε. Δεν θέλουμε ο όγκος των μεταφορών να, μειωθεί. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Εγκρός για το σχέδιο έκθεσής του παρότι ήταν άνω των 400 οι τροπολογίες, ε, κατάφερε να συγκεράσει τις απόψεις. Ευχαριστώ και τον Ζάιπα και τον συνάδελφό μου είναι η τελευταία συνεδρία στην Επιτροπή με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή στην ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑΜΟΥ. Θα ήθελα λοιπόν να του υποσχεθώ ότι θα επιδιώξουμε μία ίσως και λυμμένη πρόταση για τα δύο αυτά ζητήματα αναχείρες και ελπίζουμε να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες. Κάποια σχόλια τώρα. Οι τροπολογίες που αναγνωρίζουν την υποχρεωτικότητα του συστήματος ε, για την ε, διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ε, και την κατοχήρωση ισότιμης πρόσβασης στο τροχαίο υλικό είναι τροπολογίες που μας βρίσκουν σύμφωνες. Υπάρχει μια ομάδα τροπολογιών με τους νέους ορισμούς και πιστεύουμε ότι πραγματικά θα οδηγήσει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια κυρίως για ε, τα σχέδια δημοσίων μεταφορών για να εξασφαλίσουμε τη μη διακριτική μεταχείριση για την πρόσβαση στο τροχαίο υλικό παραδείγματος χάρη ε, μεγαλύτερη ευελιξία για τα ε, εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή τους οι τοπικές αρχές η τροπολογία 633 συνεργασία τοπικών αρχών για ομαδοποίηση τοπικών πορών τροχαίων τροχαίου υλικού, προσδιορισμός συνθήκων χρήση τροχαίου υλικού και το καθεξής. Ε, θεωρούμε ότι είναι ενδιαφέρον να συμπεριληφθεί ε, ρήτρα ε, αμοιβαιότητα. θα έπρεπε να τη διερευνήσουμε περαιτέρω. όντω η ρήτρα κυρίω κυρίως για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων θα είναι επωφελή σε σχέση με την εξωτερική ανάθεση Ε, θα έπρεπε να εφαρμόζεται αυτό και σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Αλλά φυσικά θα πρέπει να ισχύει η ημερομηνία θέση, α, ανοίγματος της αγοράς. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε όλες αυτές τις ε, τροπολογίες γιατί θα αποδυναμωθεί η αρχική μας πρόταση σε σχέση με την υποχρεωτική διεξαγωγή διαγωνισμού και φυσικά δεν μπορούμε να δεχτούμε τροπολογίε που υπερβαίνουν την αρχική μα πρόταση, όπω τροπολογίε που τροποποιούν τα ελάχιστα όρια για την άμεση ανάθεση. για τους τρόπους μεταφοράς που δεν είναι ε, σιδηροδρομικοί. να είναι απεριόριστες οι δυνατότητες εξωτερικής ανάθεσης στις υδροδρομικές μεταφορές ε, είτε θα διατηρήσουμε το άρθρο 5-6 είτε θα αποδυναμώσουμε τους όρους για την εξωτερική ανάθεση. Αυτούς τους δύο τρόπους βλέπουμε για τη μη διακριτική πρόσβαση σε βιώσιμα ε, βιώσιμο ομαδοποιημένο τροχαίο υλικό είναι το μέλλον των σιδηροδρόμων και δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε τις αρμοδιότητες σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο για να υπάρξει συμμόρφωση με τις νέες διατάξεις. Εξάλλου, οποιαδήποτε απόφαση παίρνει αρμόδια αρχή για το τροχείο υλικό δεν πρέπει να επιφέρει στρέβλωση στην αγορά. Οι όροι θέσει σε εμπορία ε, θα πρέπει να συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία της Ένωσης. Και όπως επανειλημμένα έχουμε πει, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη μεταβατική περίοδο για την υποχρεωτική διεξαγωγή διαγωνισμών στο μέτρο που αποκλίνει σε μεγάλο βαθμό από την αρχική μας πρόταση. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν με τον κύριο Τρεμόζε και σε σχέση με το ανώτατο μέγεθος το PSO δεν μπορούμε να επιλέξουμε ε, επίπεδα ε, που δεν θα επιτρέψουν ομαλή διεξαγωγή των διαγωνισμών. Είναι τόσο πολύ τροπολογίες που δεν θα μπω σε λεπτομέρειε για όλε. Θα ήταν αδύνατο να τι συζητήσουμε και Εν είδη συμπεράσματο, ε, θα έλεγα ότι ο αναθεωρημένο κανονισμό θα πρέπει να επιφέρει αναβαθμισμένε ε, υπηρεσίε ε, και χρηστότερη χρήση των δημοσίων πόρων στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι συμβαστικέ τροπολογίε που θα ψηφιστούν στην Επιτροπή Τραν, ελπιστούμε θα Τέλη Οκτωβρίου θα εξυπηρετούν αυτό το στόχο, πάντως είμαστε στη διάθεσή σας αν χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινήσεις. Ευχαριστούμε πολύ να περάσουμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Έκθεση Μπιλμπάου, Ζέλερ και Κράμερ. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μπιλμπάου. Τέσσερα λεπτά η κυρία Μπιλμπάου, Βαραντίκα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην έκθεσή μου σχολιάζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει να ε, τηρήσει τους στόχους της Λευκής Βίβλου για έναν ενιαίο άξονα μεταφορών. Υπάρχει μια κατάσταση, η οποία περιγράφω στην έκθεση, που είναι μάλλον απογοητευτική, θα μπορούσε να γίνει και απογοητευτική και καταστροφική, εάν οι διαχειριστές και τα με, κράτη-μέλη συνεχίσουν το παρόν καθεστώς και δημιουργούνται συνεχώς φραγμοί για το άνοιγμα της αγοράς και τη βελτίωση του σιδηροδρομικού τομέα. Θα ήθελα να σας ζητήσω κύριε Πρόεδρε να γίνει λίγο ησυχία διότι πραγματικά αποσυντονίζομαι, ακούω ότι όλο τον κόσμο μιλάει από όλες τις πλευρές. Σας παρακαλώ όσοι θέλετε να αποχωρήσετε από την αίθουση, σας παρακαλώ να αποχωρείτε ησύχω, αλλά με εκπλήσει που θέλει να φύγει κάποιο τη στιγμή που συζητάμε τη διαλειτουργικότητα, αλλά τέλος πάντων. Κύριε Μπιλμπάου, λοιπόν, θα υπάρξουν οι εντάσεις. Ε, υπάρχει ανάγκη να διαχειριστεί το καθεστώ, να παραμείνει το καθεστώς, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχει ο κατακαιρματισμός, ο διαχωρισμός, το κόστος ε, το οποίο θα είναι αυξημένο για τους κατασκευαστές σιδηροδρομικών οχημάτων και θα υπάρχει αυτή τη στιγμή όπως έχει κατάσταση ε, για το κατασκευαστή ενός οχήματος μπορεί να στοιχήσει και μέχρι 6 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να διαρκέσει και δύο χρόνια η όλη διαδικασία για την έκδοση αδειών σε διοικητικό επίπεδο. Αυτό που θέλουμε είναι να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση και φαίνεται ότι ω προς τη διάγνωση τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια διάγνωση για το τι γίνεται με την τρίτη δέσμη μέτρων και να μπορέσουμε τουλάχιστον να έχουμε πολιτική βούληση ώστε τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα τηρήσει τους όρους αυτής της τρίτης δέσμης να τα προχωρήσουν και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στη συνέχεια. Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία θηρίδα και θα πρέπει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός να μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη των ε, εθνικών συστημάτων και να μπορεί να βοηθήσουν και οι εθνικές αντίστοιχες υπηρεσίες. Για να μπορέσουμε επίσης να έχουμε εθνική μεγαλύτερη διαφάνεια και να υπάρχει και ανταγωνισμό στο θέμα των σιδηροδρομικών μεταφορών, θα μπορούσαμε ίσως να βελτιώσουμε μέσω των προτάσεών μας τη διαφάνεια ε, οι επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα και όλο το κόστος και τα κονδύλια τα οποία δίνονται τώρα για τις διοικητικές διαδικασίες και τις καθυστερήσεις να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουμε ασφάλεια δικαίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι διατεθειμένες να επενδύσουν στον τομέα και να είμαστε υπέρ καινοτομίας ώστε οι μεταφορές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποτελούν και σημεία αναφοράς παγκοσμίως. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι η στόχη. Ε, 440 τροπολογίες υπευλήθησαν. Δεν θα κάτσω φυσικά τώρα να τις σχολιάσω όλες, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν δύο ουσιαστικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε και από αυτές τις 440 ε, τροπολογίες νομίζω ότι διαφαίνονται σαφώς. Εμείς είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων να έχουμε μία ενιαία ε, μεταχείριση που θα επιτρέπει να εκδίδονται όλες οι άδειες ε, από την ίδια αρχή και ζητήσαμε μια μεταβατική περίοδο 5 ετών ώστε αυτή η μετάβαση να γίνει και με τη βοήθεια των αρμοδίων αρχών σε εθνικό επίπεδο. Διότι ε, είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Αεροπορία μπόρεσε να κάνει αυτή τη μετάβαση και θα ήθελα να σας δώσω το εξή στοιχείο. Εδώ στην Επιτροπή πολύ συχνά ακούμε πολλούς ευρωβουλευτές να λένε ότι είναι αδύνατο να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και γιατί αυτό βιώνουμε κρίση και δεν έχουμε κατάλληλο προπολογισμό. Πρέπει να πω ότι μετά από τη συνεδρίαση που κάναμε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό πραγματικά βρέθηκα προ μια ευχάριστη ε, εκπλήξεως διότι μας είπαν ότι δεν στοιχίζει τίποτα για τον ε, δημόσιο καβανά μπορούν ε, να καλύψουν αυτοί, κερδίζουν χρήματα από τις εργασίες τους και έτσι υπάρχει οικονομική δυνατότητα να προσφέρεται αυτή η υπηρεσία. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε. Ποιος είναι ο ρόλος ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και των Εθνικών Οργανισμών και τι θα πρέπει να γίνει και πώς ε, θα πρέπει να διαχειριστούμε τα ξεχωριστά αυτά δίκτυα, εάν πραγματικά υπάρχουν δίκτυα τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε αυτή τη διαφορετική κατάσταση. Κατά τα λοιπά νομίζω ότι είναι σαφή τα πράγματα και θα μπορούσαμε να έχουμε ε, συμφωνία για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ κύριο Σαλκαντράου για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια εκ μέρους της Ινίσα Αγία Σάντερ της Κιώδης εισηγητριός μας που δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Έχουμε καταθέσει αρκετές τροπολογίες, καταρχάς ως προς το πεδίο εφαρμογής. Έχουμε καταθέσει μία ε, τροπολογία για να μπορούν να έχουν συστήματα ελαφρών τρένων, όπως για παράδειγμα τύπου μετρό αν το επιθυμούν. Ε, αυτή είναι αλλαγή που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ε, ε, προτείνει αλλαγή των προδιαγραφών, αλλά επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προ το παρόν είναι θελοντικό, θα θέλαμε να παραμείνει. Δεν θέλουμε να αποκλείουμε τι τοπικέ υπηρεσίε και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ε, καθορίζουμε συγκεκριμένε εξαιρήσει. Όσον αφορά την κινητικότητα, έχουμε καταθέσει αρκετέ τροπολογίε για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των υπευθύνων αρχών όταν θα καταρτήσουμε το σχέδιο και επίσης δεν θα πρέπει να γίνεται περαιτέρω επαλήθευση για την ίδια περιοχή με τις ίδιες τεχνικές ε, απαιτήσεις. Θα μπορούσε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και τις δεξιότητές μας εάν οι κατασκευαστές και οι, ε, οι διαχειριστές μπορούν να έχουν το ίδιο υλικό το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται παντού και να είναι και έτσι αρκετά ανταγωνιστικό. Ως προς το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του TSA θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι θα μπορεί να γίνει αυτό αν υπάρχει κατάλληλη εκτίμηση που αναλύει το κόστος και τι θα γίνει με την εφαρμογή και τα αναμενόμενα ωφέλη και για τους ε, οικονομικούς φορείς και για τους διαχειριστές. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ των τρένων ε, ε, μεγάλης ταχύτητας και των συμβατικών τρένων, διότι τα τρένα μεγάλης ταχύτητας ε, λαμβάνουν πολύ σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά και επιπλέον στοιχεία και επομένω υπάρχει διαφορά σε σχέση με το συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Για οχήματα τώρα τα οποία έχουν χαμηλή κατανάλωση άνθρακα γνωρίζετε ότι υπάρχει διαφορά στα εμπορικά βαγιόνια στην Ευρώπη. Αυτό ίσως θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένες αμαξοστοιχίες οι οποίες ε, δεν είναι σχεδιασμένες για να μεταφέρουν εμπορεύματα. Η κυρία Γιάλα προσπαθεί να διευκρινίσει ε, κάποια στοιχεία και θέλει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τομέα. Τέλος, για το RTMS Θεωρούμε ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός θα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο, αλλά ο ρόλος των εθνικών ε, οργανισμών θα πρέπει να είναι σημαντικός, γιατί αυτοί γνωρίζουν καλύτερα πώς έχει η κατάσταση, για να ε, βελτιώσουν, ότι τα, να ελέγξουν συγγνώμη, τα συστήματα RTMS δεν έχουν προβλήματα σε σχέση με τα συμβατικά δίκτυα. Αυτά λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα των τροπολογιών που κατέθεσε η σκιώδης συγγητρία μας και ε, θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στην εισηγήτρια και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ, να ευχαριστήσω τον εισηγήτη. Την εισηγήτρια μάλλον, γιατί έχουμε πολύ καλή ε, συνεργασία και η πρόταση αποτελεί μια πολύ καλή βάση. Ε, έχει, έχει υπάρξει μεγάλη υποστήριξη για τις τροπολογίες. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες ε, για το διαχωρισμό μεταξύ της ε, ε, έγκρισης των διαφόρων επιχειρήσεων που, θα πρέπει να, που σημαίνει ότι θα μπορούν τα τρένα να αγοράζονται μετά από έγκριση. Μόνο τα εγκεκριμένα μάλλον και τα τεχνικά τεστ θα μπορούν να γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αδειοδότησης ευρωπαϊκό. Η Κομισιόν μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα, ενώ το έχει αποφασίσει εδώ και κάποιο καιρό. Ε, Επίση, το Ευρωπαϊκό Μητρό χρειαζόμαστε και το υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε να γίνει Ευρωπαϊκό Μητρό. Πρέπει βεβαίω να υπάρξει δυνατότητα ενίσχυση των ανθρώπων με μειωμένη κινητικότητα. Και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι όσοι δεν το χρειαζόμαστε, αλλά για αυτού που το χρειάζονται θα πρέπει να προνούμε να του δώσουμε τι απαραίτητε ε, υπηρεσίε. Μετά, Έχουμε 6.000 RTMS ε, ε, χιλιόμετρα στην ε, Ευρώπη και δεν μπορεί να ταξιδέψει κανένα όχημα πάνω σε αυτά. Αυτό πρέπει να διορθωθεί άμεσα γιατί αλλιώ θα έχουμε την ίδια καταστροφική κατάσταση με πάρα πολλέ επενδύσει που έχουν γίνει. Πρέπει επίση να υπάρξει ρύθμιση για την, ε, ε, για την NSA και την ERA. Ε, Βεβαίω η ERA βεβαίως δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή δεν μπορεί να ρυθμίσει τα πάντα που κάνουν οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει στο μέλλον να προχωρήσουμε με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με, την ευρωπαϊκή, ε, με μια ευρωπαϊκή, ένα ευρωπαϊκό ενιαίο πρόγραμμα. Επίσης, συνεργασία μεταξύ των εθνικών και της ευρωπαϊκής αρχής, ε, αριθμιστικής αρχής. Το Συμβούλιο έχει ε, υποβάλει έναν συμβιβασμό. Είναι ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πάει όσο μακριά πρέπει. Λέει ότι οποιοδήποτε τρένο ταξιδεύει στην Ευρώπη θα το αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή. Αλλά τι, τι ακριβώς πιστεύει ότι γίνεται στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους το Συμβούλιο. Ας πούμε, Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία. Με βάση το, τα όσα έγιναν στο παρελθόν έχουν ένα παλιό σιδηροδρομικό δίκτυο. Παρ' όλα αυτά, σήμερα δεν υπάρχει ε, τρένο που να πηγαίνει από, την, ε, από το Ταλίν στη Ρήγα, ας πούμε. Πρέπει να υπάρξουν ε, μετεπιβιβάσεις κτλ. Ε, προφανώς αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Στη Γαλλία τώρα έχουμε ένα ενιαίο κράτος, αλλά έχουν διαφορετικά συστήματα σιδηροδρομικά μεταξύ Βόρειας και Νότιας Γαλλίας. Αυτά είναι γελία πράγματα. Γι' αυτό αυτή η προσέγγιση είναι, ενισχύει την εθνικιστική οπτική. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή οπτική. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν, να συνεχίσουν οι διάφορε δραστηριότητε που υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ζήλε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Ήταν πολύ καλή συνεργασία μας, κυρίω για τον τεχνικό πυλώνα. Ε, θα βασιστώ στα σχόλια του Μάικλ. Ε, μπορείς να πας από, τη, ε, το Βίλνου στη Ρίγα και στο Τάλιν μέσω των, τεν, ε, της, των ευρωπαϊκών δικτύων. Ε, θα συμφωνήσω ότι δεν είναι πολύ καλή η διασύνδεση, αλλά... Δεν μπορούμε να σταματήσουμε στη διαπίστευση των οχημάτων. Το θέμα είναι ότι είναι μεγάλες οι αποστάσεις και είναι πολύ χαμηλή η ταχύτητα και άρα η εμπορική αξία δεν είναι αρκετά υψηλή και 10 ε, ε, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πρόσφατα των τέντη. Ε, για τη διαλειτουργικότητα τώρα, αυτό συνδέεται και με τις απομονωμένες χώρες. Υπάρχουν δύο ομάδες απομονωμένων δικτύων κατά τη γνώμη και γι' αυτό κατέθεσα και αυτή την τροπολογία για να εξευρεθεί μια καλή συμβαστική ε, τροπολογία. Υπάρχουν λοιπόν απομονωμένα δίκτυα στην Ευρώπη και σε άλλες τρεις χώρες υπάρχουν, ε, σε τρεις χώρες, συγγνώμη, σε τρίτες χώρες υπάρχουν άλλα ολοκληρωμένα ε, δίκτυα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις. Αν θέλετε τώρα να τιμωρήσουμε κάποιους φορείς, κάποιους παίχτες αγοράς ε, που επιδιώκουν αδειοδότης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις φωνές ε, τρίτων χωρών που μας παρακαλούν να μην δίνουμε συγκριτικό πλεονέκτημα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εάν εγκρίνουμε το νομοθέτημα ως έχει θα έχουμε εμπορικό ε, πόλεμο. Ας μην το ξεχνάμε, αν, παραμείνει, αν έχουν οι διατάξει για το RTMS, έχουμε πολλές ε, τροπολογίες ε, που μας μιλάνε για, τα, για τους συμβατικούς σιδηροδρόμους και για τα παρατρόχια συστήματα ελέγχου και χειρισμού. Θα πρέπει όμως να δούμε ολοκληρωμένα το ζήτημα και σε συνδυασμό με αυτό του ευρωπαϊκού μητρώου οχημόταν γιατί χρειαζόμαστε ολοκλήρωση και με τα συστήματα τρίτων χωρών. Τι θα γίνει με το τροχαίο υλικό ε, και τα οχήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, παραδείγματος χάρη, δεν έχουν τις κατάλληλες βάσεις δεδομένων. Είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο γιατί πήγαμε, τα επισκεφτήκαμε, τα είδαμε. Δεν υπάρχουν υπάρχει Παραδείγματο χάρη στη Φινλανδία, ε, συμβατό τροχαίο υλικό. Καταλαβαίνετε, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστούμε, Κόλιτσετ. <laughs> Tak, děkuji. Já bych eh, několik poznámeček. Sjednocení technických požadavků a certifikačních. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για την ε, όλη αυτή διαδικασία αδειοδότησης και για τις ενιαίες διατάξεις ε, νομίζω ότι είναι σωστά και είναι το ουσιαστικό. Ε, τα υπόλοιπα που συζητούμε οδηγούν ίσως σε πιο δυσχερή κατάσταση του σιδηροδρόμου. Είναι σημαντικό να υπάρξει μία ενιαία πιστοποίηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγνωρίζεται και δεν μιλούμε ε, μόνο για τα ομιτρό, μιλούμε για όλα τα είδη πιστοποίησης ε, των ε, δικτύων. Καλό θα ήταν να έχουμε πιστοποιημένα οχήματα. και θα πρέπει να έχουμε και μια ενιαία διαδικασία για όλα αυτά. Επίσης, οι τεχνικές απαιτήσει, αλλά και οι διαδικασίες είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή από κοινού με τις εθνικές αρχές θα πρέπει να το μελετήσει. Ε, αντί να έχουμε 26 διαφορετικά εθνικά συστήματα με 26 διαφορετικά σετ απαιτήσεων, να έχουμε ένα θα πρέπει όντω να υπάρξουν αυτά τα νέα πιστοποιητικά μαζί με την ε, όλη η διαδικασία την ελεκτική που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την όλη διαδικασία. Βεβαίως υπάρχουν κάποια κομμάτια του σιδηροδρόμου που είναι απομονωμένα ε, ή που δεν, που δεν έχουν το σωστό εύρος. Όντω ε, οι χώρε τη Βαλτική είναι μια ειδική περίπτωση, αλλά νομίζω ότι ε, είναι λίγο νωρί να μιλούμε για νέε διατάξεις για εκεί. Η κυρία Στέλλας νομίζω θα πάρει το λόγο για να ε, εκπροσωπήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Ήθελα να ακούσω πρώτα τον να μιλήσω συγγνώμη εξ του κύριου Γκράντες Πασκουάλ, ο οποίο δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα και μου έδωσε αυτό το σημείωμα, το οποίο καθόρισε με του συντονιστέ για την οδηγία για τη βιολετουργικότητα και περιλαμβάνει και τι 29 τροπολογίες που υπευλήθησαν στην ε, πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν ε, σας πω για τη θέση μας, θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μεταρρύθμιση του τρίτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους και γι' αυτό ακριβώς είχαμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ίσως δεν είναι τόσο φιλόδοξη ή είναι περισσότερο φιλόδοξη λόγω των τροπολογιών που υπευλήθησαν. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά διαλεκτουργικό δίκτυο για τους σιδηροδρόμους για όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ακριβώς και συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγήτρια της ε, έκθεσης και πολλές από τις τροπολογίες της και θεωρούμε ότι όλο το σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε μια βαθμιδόν εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων με πολύ σαφείς προθεσμίες οι οποίες ε, θα βοηθούν να γίνονται οι μεταρρυθμίσεις και να είναι συμβατές με τα συστήματα τα οποία λειτουργούν σωστά αυτή τη στιγμή. Υποστηρίζουμε λοιπόν το προστιθέμενο όφελο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε υποβάλει αρκετές τροπολογίες οι οποίες συνοψίζουν τη θέση μας και συνάδει και με τη θέση άλλων ε, πολιτικών ομάδων και θεωρώ ότι θα δώσει και το έναυσμα για συμφωνίες στο μέλλον. Η τροπολογία για την έγκριση των... Ε, και διάθεση στην αγορά συνδυροδρομικών οχημάτων είναι το πιο σημαντικό. Θέλουμε να διευρύνουμε ε, τη δυνατότητα ε, κυκλοφορίας διαφόρων σιδηροδρομικών οχημάτων και θεωρούμε ότι όπως ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δυσχεραίνεται η χρήση συγκεκριμένων οροχημάτων όταν βρίσκονται σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές ε, αρχές ασφαλείας βάσει της ε, ευθύνης τους ε, όταν υπάρχει και κατάλληλο αίτημα να δίνεται έγκριση για τη διάθεση στην αγορά ενός οχήματος όταν πρόκειται για οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε μια περιορισμένη περιοχή, σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο το οποίο βρίσκεται σε ένα μόνο κράτος μέλος. Επιπλέον, οι 8 ε, τροπολογίε οι οποίε υπευλήθηκαν για το άρθρο 8 ε, συνοψίζουν και κάποιο άλλα στοιχεία τα οποία αφορούν τη ε, συμβιβασμό μα Το να υπάρχουν, ε, για παράδειγμα, σταθερές υποδομές, αυτές θα καθορίζονται από τις εθνικές αρχές κατά την άποψή μα, διότι μέχρι τώρα ήταν επιτυχής η διαδικασία. Θα μπορεί να υπάρχει βέβαια δυνατότητα διαβούλευση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων και να μπορούν να λαμβάνει υπόψη η γνωμοδότησή της ε, πριν από την έγκριση, ώστε το RTMS να έχει κάποια συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι το σύνολο των προτάσεων και για τη δέσμη μέτρων των σιδηροδρόμων ήταν πολύ πολύ και γι' αυτό ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγήτρια διότι θεωρούμε ότι αυξάνει την προστιθέμενη αυξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδίδει μεγαλύτερη ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές, ε, καλύτερες δυνατότητες ε, ανταγωνισμού και την πραγματική πρόταση για αποτελεσματική διαλειτουργικότητα. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο ε, στον κύριο Κράμερ για τη δική του έκθεση, που είναι η έκθεση για τον ε, τομέα των σιδηροδρόμων αναδιατύπωση. Τέσσερα λεπτά. Ναι, να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συζητητές. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας. Και αν δούμε τις 426 ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, είναι κυρίως συμπληρωματικές στο κείμενο. Έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, έχουμε ευρωπαϊκή οπτική για την ασφάλεια, δεν έχουμε μεγάλε διαφορέ στι απόψει μα. Χαίρομαι ιδιαίτερω για την υποστήριξη για την εισαγωγή ενό ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ασφαλεία, ότι οι εθνικοί ε, κανόνε θα πρέπει να ενοποιηθούν υπό την ε, αιγίδα τη Ευρωπαϊκή Αρχή, ότι θα υπάρξει συντονισμό. Υπάρχουν 12.000 ε, κανόνε τώρα, κάθε κράτο φτιάχνει του δικού του. Θα πρέπει λοιπόν να απαλείψουμε πάρα πολλούς. Ε, ε, υπάρχουν τόσοι γραπτοί και άλλοι τόσοι ε, προφορικοί κανόνες. Όλα αυτά είναι τρελά. Πρέπει να υπάρξει λίγο ρεαλισμό στην Ευρώπη. Τώρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το θέμα της των εργαζόμενων στην ασφάλεια, τον χρόνο ξεκούρασής τους, τον, τις ώρες που θα εργάζονται. Πρέπει να ε, Βεβαίω για του σιδηροδρόμου οι συνθήκε είναι λίγο καλύτερε από ότι για τι αεροπορικέ μεταφορέ. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρξει καλύτερη συντονισμό. Ε, Επίση για του κινδύνου που διατρέχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε. Η πρακτική στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δείξει που υπάρχουν προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρξει Εμπιστοσύνη λοιπόν και καλή ε, εκπαίδευση ώστε να αποτρέπονται τα ε, ατυχήματα. Επίσης ε, τα πρότυπα για τον θόρυβο πάντα βεβαίω αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια αλλά και για τη συντήρηση έχουν υπάρξει πολλά δυστυχήματα που συνήθως δεν φταίνε τα, τα οχήματα, φταίνε συνήθως τα ελληπή πρότυπα στο Βερολίνο έχουν υπάρξει κάποιε τέτοιε περιπτώσει ε, δυστυχημάτων που οφείλονται σε λυπή πρότυπα ασφάλεια, οπότε αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα. Οι εξαιρέσει τώρα για τι τοπικέ ε, και περιφερειακέ αρχέ ε, θα πρέπει να περιοριστούν πολύ προσεκτικά. Εγώ είμαι υπέρ να μην ε, υπάρξει ένα σύστημα για όλες τις ε, χώρες, ε, να υπάρχουν κάποιες μεν εξαιρέσεις, αλλά όπως είπα η εθνική, η οπτική είναι λαθασμένη. Πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή. Ίσως όμως για κάποιες περιφέρειες να είναι δυνατό να μην υπάρχει ευρωπαϊκή ενοποίηση των κανόνων. Μετά πρέπει να έχουμε μια σύντομη συμφωνία. Συμφωνήσαμε, ήμασταν όλοι ως προς αυτό θετικοί. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα συμβασμός με το Συμβούλιο και χάρη στη συμφωνία του Συμβουλίου φτάσαμε ένα βήμα παραπέρα. Την προηγούμενη Πέμπτη η Γερμανία ευτυχώς πιέστηκε και μετακινήθηκε προς την ε, ε, σωστή κατεύθυνση. Ε, ο συμβασμός βεβαίως είναι ε, μισό βήμα προς τα εμπρός. Θέλουμε να πάμε πιο μπροστά. Δεν θέλουμε να υπάρξουν διαμάχες μεταξύ των εθνικών και της Ευρωπαϊκής Δεθμιστικής Αρχής. Θέλουμε να υπάρχει καλή συνεργασία και πρέπει, πρέπει να συνεργάζονται καλά οι αρχές αυτές με την Ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή Αρχή μπορεί να έχει τον τελευταίο λόγο, έτσι ώστε να υπάρξει ο θεμέλιος λίθος για εναρμόνιση στο μέλλον. Ξέρουμε ότι είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία αυτή. Το είδαμε και για τι αεροπορικές μεταφορές, Κάναμε πολλές ε, συζητήσεις και με τους συγητέ, αλλά ήταν πολύ επικοδομητικές. Και τι έγινε βέβαια τελικά. Σήμερα Χαιρόμαστε που έχουμε λύσει τα προβλήματα. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τους, για τους σιδηροδρόμους. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, εξασφαλίσουμε και να εξυπηρετήσουμε και τους επιβάτες, να μπορούμε να τους, παράχουμε, να τους παράσουμε περισσότερες υπηρεσίες με λιγότερα ή τουλάχιστον με τα ίδια χρήματα. Ευχαριστώ κύριο Δεμπακ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάχ ε, μου ζήτησε να μιλήσω εγώ εκ μέρους του. Ε, Βεβαίω θέλουμε να υπάρξει ασφάλεια στα πλαίσια του τέταρτου πακέτου για του υδροδρόμου. Θέλουμε να υπάρχει βεβαίω αυτή σε συνάφεια και με τα υπόλοιπα κομμάτια του πακέτου. Η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή είναι σημαντική. Η διαλειτουργικότητα επίση και πρέπει να την έχουμε υπόψη. Ιδιαίτερο σημαντικό είναι για την ευρωπαϊκή, να τονίσουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ο στόχο είναι να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αρχή και να έχουμε και το ενιαίο επιστοποιητικό ασφάλεια, έτσι ώστε να υπάρξει ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Μόνο έτσι στο τέλος θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη ασφάλεια στους υδροδρόμους και λιγότερο κόστος καθώς και θα μπορούμε να μειώσουμε τους χρόνους. Αυτό που προτείνει ο εισηγητής ε, νομίζω ότι ε, αναφέρονται και στις περισσότερες ε, τροπολογίες που έχουν, που έχουν υποβληθεί. Έχουν υπάρξει κάποιε τροπολογίε από το ΕΛΚ, δεν θέλω να τι ε, αναφέρω. Ε, τα βασικά σημεία για μένα είναι ε, ότι πρέπει να υπάρχει σαφή ορισμό των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων και σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα κενά. Δεύτερον, περισσότερη προσοχή στην συντήρηση. Εδώ μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να μιλήσουμε για την διατήρηση, για την καλύτερη συντήρηση του τροχαίου υλικού και των οχημάτων. Τρίτον, τα κοινωνικά, οι κοινωνικέ πτυχές, ε, το, τα ωράρια εργασίας, οι ε, ώρα ξεκούραση είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τονιστούν στην έκθεση. Ε, τέταρτον, σε αυτή την κατηγορία πρέπει να υπάρξει όντως σωστή νοοτροπία, το είπε και ο εισηγητής. Το είχαμε κάνει πριν από λίγα χρόνια και για τις αεροπορικές μεταφορές. Ε, οι υπάλληλοι ας πούμε, που έχουν κάνει λάθη ή έχουν ανακαλύψει κάποια κενά ασφάλεια θα πρέπει να μπορούν να τα δηλώσουν χωρί να φοβούνται ότι επειδή δήλωσαν κάποιο κενό ασφάλεια θα χάσουν τη ζωή του. Ο κύριο Μπαχ ε, εύχεται στον εισηγητή καλή τύχη και ό,τι καλύτερο για να υπάρξει συμφωνία για την έκθεσή του. Ευχαριστώ. τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Η Ένες Αλαγιάλα Σέντερ είναι η μας και εξ ονόματός της θα ήθελα να εξηγήσω λίγο τις τροπολογίες που καταθέσαμε και να μιλήσω και για διάφορες τροπολογίες που απηχούν την Ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ατυχήματα στην ε, ε, αεροπορία, στην πολιτική αεροπορία με αντιστοιχεία για τους σιδηροδρόμους. Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε δεδομένα για τους, εργοδηγούς, για τους ε, μηχανοδηγούς και για τα δίκτυα για να ενισχύσουμε την ασφάλεια. Μιλάμε για την έννοια της fair culture, ούτως ώστε το προσωπικό να ενθαρρύνεται να καταγγέλει περιστατικά ασφαλείας. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα ατύχημα, το πρόβλημα είναι ο εντοπισμός των θυμάτων. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει ε, μέρες ολόκληρες, όπως είδαμε και το καλοκαίρι στην Ισπανία και γι' αυτό βάλαμε μια Λογική σκέψη και καλούμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμου να προβλέψει την εναλλακτική να υπάρχουν τα ονόματα των επιβατών στι ε, γραμμέ ε, υψηλή ταχύτητα στην Ισπανία και στη Γαλλία, όπου είναι υποχρεωτική η κράτηση, παραδείγματο χάρη, και έχουν τόσο ή άλλω τα ονόματα των επιβατών. Θα θέλαμε επίσης να ενισχύσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα που εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο. Ένα... Θα πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω την προσέγγιση που βασίζεται προς το παρόν μόνο στα συστήματα. Για την αναβάθμιση της ασφάλειας στην Ένωση προτείνουμε να έχουμε ε, ένα σύστημα πλεονάζοντος προσωπικού σε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην εξαρτώμεθα από ένα μόνο σύστημα. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τώρα ε, τόσο ε, οι εθνικές αρχές όσο και διαχειριστές υποδομών όσο και η παροχή θα πρέπει να έχουν σχέδια πρόσβασης και αρρωγής σε περίπτωση ατυχήματος, ένα σχέδιο για την περίθαλψη των θυμάτων και ένα γενικότερο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Και αυτά πιστεύουμε ε, και γι' αυτό ε, το αναφέρω και στη δική μου την έκθεση, ότι ο διαχειριστής υποδομής σε διασυνοριακό επίπεδο θα πρέπει να έχει ένα συντονιστικό σχέδιο για διαχείριση σε περίπτωση ατυχήματος, ούτως ώστε να μπορέσει σε περίπτωση ατυχήματος να υπάρξει αυτή η διασυνοριακή συνεργασία. Σαφής πρέπει να είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα στις συμβατικές ε, και τις υψηλής ταχύτητας γραμμές και για τη συντήρηση έχουμε την ελάχιστη συντήρηση για τα οχήματα και πρέπει να προσαρμόσουμε τα κριτήρια ε, ως προς ε, το είδος ε, τροχιάς, το είδος οχήματος και να μην λαμβάνονται υπόψη μόνο οι χιλιομετρικές αποστάσεις που έχει κάνει κάθε όχημα για το χρόνο εργασίας και ανάπαυσης ε, των οδηγών. Έχουμε καταθέσει επίσης τροπολογίες. Κατά τα άλλα συμφωνούμε με την εισηγήτρια κυρία Μπιλμπά. Ευχαριστούμε. Μπαίνει τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Ναι, έχω καταθέσει διάφορες τροπολογίες για να τονίσω τη σημασία που έχει η έννοια του reasonably practicable, όπως λέμε στα αγγλικά πρέπει να αποδείξουμε ότι το κόστος που επισύρει η μείωση του κόστους δεν είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το κέρδος, το αποκτηθέν κέρδος έχουμε πολλούς απόλυτους παράγοντες ε, στο, στον τομέα της ασφάλειας, αλλά τι θα κάνουμε, αν συνεχίσουμε έτσι θα πρέπει να αποκλείσουμε τους σιδηροδρόμους, γιατί δεν είναι ανταγωνιστική εμπορική πρόταση που κάνουμε. Δεύτερον, για την απόδοση ευθυνών πρέπει να προσέξουμε όταν λέμε ότι όλοι φέρνουν την ευθύνη, όλοι οι φορείς. Ναι, είναι, αλλά ε, ευθύνονται για το δικό τους κομμάτι μέσα από τις ε, συμβατικές τους υποχρεώσεις. Δεν θέλουμε να υπάρξει σύγχυση, κυρίως για τον ε, πελάτη. Ο πελάτης έχει σύμβαση με τον προμηθευτή με την επιχείρηση δηλαδή και όχι με την φορτωτική ή οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται στην αλυσίδα. Εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα ενίο σημείο για να αποτείνεται ο πελάτης σε περίπτωση προβλήματος. Τώρα για τις τροπολογίες που επιτρέπουν τα κράτη-μέλη να ε, εισαγάγουν υψηλότερες προδιαγραφές ε, ασφαλείας. Σε περισσότερες περιπτώσεις δεν θα τεθεί ζήτημα διαλειτουργικότητας ε, για τη δημιουργία του ενιαίου χώρου, σιδηροδρομικού χώρου, αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και να ακολουθούμε αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν ναι, με να έχουμε υψηλέ προδιαγραφέ ε, ασφαλεία, αλλά όχι ει βάρο τη εναρμόνιση. Εάν αυτό συμβαίνει, θα χρειαστεί να ξαναρχίσουμε και σε μία δεκαετία από τώρα ε, θα, έχουμε, ε, θα έχει επικρατήσει ένα πλήρες χάος και θα είναι κατακαιρματισμένη η αγορά. Για τις ώρες εργασίας δεν πρέπει να ζητήσουμε ε, νομοθετική ρύθμιση για αυτό το ζήτημα, να ασχοληθούμε μόνο με την ασφάλεια. Είδαμε και τον φλεγόμενο περιστατικό της περασμένης εβδομάδας, αλλά δεν θα έπρεπε τώρα κοινωνικά ζητήματα να συμπεριληφθούν σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε, Τζίλερ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τον Μάικλ για την τόσο καλή συνεργασία που κάνουμε για τον τεχνικό πυλώνα. Είπατε ότι οι γερμανικές αρχές συμφωνούν και ότι θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε εναρμόνιση και στα τεχνικά ζητήματα. Βέβαια, νομίζω ότι θα διήστανται και απόψε εδώ στην Επιτροπή μας, πέρα από τις εθνικές απόψεις. Θα, δει, θα δούμε. Για τα ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας, ο Μιχαήλ έκανε πολύ καλή συνεδρίαση με τους κοιόδης και πήραμε την εμπειρία που είχαμε από την πολιτική αεροπορία για να δούμε τι μπορούμε να διδαχθούμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, για την ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία και να τα μεταφέρουμε ε, στα θέματα ασφαλείας των σιδηροδρόμων. Ε, δεν έχουμε όμως ενιαίο τέτοιο πιστοποιητικό στην αεροπορία. Εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα των εθνικών αροχών. Ορισμένες φορές υπάρχει ένας πάροχος που θέλει να δραστηριοποιηθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος και τότε πρέπει να δούμε αν η εκεί αρμόδια εθνική αρχή μπορεί να εκδώσει αυτό το πιστοποιητικό και να δούμε, να μεριμνήσουμε ώστε να ε, υπάρχει συνοχή, γιατί σας είπα για τα συστήματα ελέγχου χειρισμού και σηματοδότησης, για τα παρατρόχια δηλαδή συστήματα, βλέπουμε ότι οι τροπολογίες των μελών της Επιτροπής ε, τα αφήνουν όλα στο RTMS. Το RTMS όμως πρέπει να συνδέεται με τις ε, ε, τοπικές αρχές. Ε, δηλαδή δεν μπορούμε να υιοθετούμε αφενός ευρύτερη προσέγγιση για κάποια ζητήματα και αφετέρου να τα αφήνουμε όλα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων γιατί πρέπει να είμαστε και ανταγωνιστικοί και υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα ε, διαλειτουργικότητας. Ελπίζουμε η τελική λύση να μην είναι αμφιλεγόμενη και να συμφωνήσουμε. Ευχαριστούμε. Κόλλητσεκ τρία λεπτά. Pokrývá do určité míry podobné, podobnou plochu jako ta zpráva předchozí. Je tady navíc. Αυτή η έκθεση δημιουργεί τρόπον την τα ίδια προβλήματα όπως και προηγούμενες. Ετίθεται και ζητήματα όπως ε, τα ωράρια ε, εργασίας. Αυτά ε, τα προβλήματα έχουμε αντιμετωπίσει και στον τομέα της αεροπορίας. Και όπως και οι οδικές μεταφορές τώρα τίθενται και στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Εγώ θα συμφωνήσω με τον ομιλητή που μας λέει ότι ουσιαστικά ε, πρέπει να βασιστούμε στα γεγονότα για να προτείνουμε μία λύση. Χρειαζόμαστε μία ομοιόμορφη διαδικασία όπου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιδροδρόμων θα φέρει την ευθύνη. Θα γίνονται σχετικές, τα σχετικά τεστ, σχετικές δοκιμές και βεβαίως θα υπάρχουν και οι δυνατότητες συντήρησης. Τώρα, σε αντίθεση με, την, με τις αεροπορικές μεταφορές, εδώ πρέπει να κάνουμε ελέγχους στις υποδομές και συντήρηση, γιατί οι υποδομίες είναι ουσιώδεις για την λειτουργία του όλου συστήματος. Αυτά από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Ε, νομίζω ότι είναι σαφής η θέση και αυτού και η δική μου. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Ζήλε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που κατέθεσαν 408 τροπολογίες στο θέμα αυτό και να πω ότι ένα σημαντικό στοιχείο είναι, σημαντικό τμήμα των τροπολογιών μάλλον, είναι τεχνικές και διευκρινιστικές, τις οποίες δεν έχω κανένα πρόβλημα να δεχτώ και να συμπεριλάβω. Άλλο τμήμα των ε, τροπολογιών είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, αλλά δεν είναι πολύ διαφιλονικούμενα και ευαίσθητα. Υπάρχει για παράδειγμα μια ομάδα τροπολογιών που αφορούν το όχι μόνο την έκδοση αδειών αλλά την ανανέωση, την αναστολή λοιπά αυτού του ενιαίου πιστοποιητικού. Ε, αν αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο εθνικό για κάποιον διαχειριστή σε εθνικό επίπεδο θα δούμε πώς θα γίνει και θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες εδώ. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Για τις συστάσεις τώρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων υπάρχουν πολλές ε, τροπολογίες για το θέμα αυτό και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο καλό συμβιβασμό από αυτού. Όσον αφορά τώρα τις προθεσμίες ε, και τις εφέσεις υπάρχουν πάλι κάποιες ομάδες τροπολογιών και εδώ νομίζω μπορούμε να βρούμε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις. Υπάρχει μια τροπολογία για το επίπεδο των τελών και των χρεώσεων που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να διαφοροποιήσουμε και τις χρεώσεις ανάλογα με την ε, ε, ε, περιοχή στην οποία υπάρχει το συγκεκριμένο σιδηροδρομικό δίκτυο. Θα πρέπει να την εξετάσουμε αυτή την πρόταση και να πρέπει να κατανοήσουμε ίσως ότι δεν είναι όλη η ίδια η αγορά και ορισμένες φορές ε, οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες για γλωσσικούς λόγους δεν αντιλήφθηκα κάποιες από τις τροπολογίες όταν θα μεταφραστούν ίσως ε, για τα θέματα μετάφρασης των πιστοποιητικών στις επίσημες γλώσσες κλπ. Ε, ε, εάν είναι γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια επίσημη γλώσσα, διότι υπάρχουν κάποιες περιοχές τις οποίες δεν χρησιμοποιείται επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο από νομική σκοπιά για μένα είναι λίγο ε, αδιανόητο. Κάποιες μη ευρωπαϊκές γλώσσες εξακολουθούν να είναι έγκυρες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας. Για μένα είναι σχεδόν παράνομο αυτό. Και τέλος, να πω ότι πρέπει να κατανοήσουμε καλά τι γίνεται με το θέμα της υπεργολοβίας των εθνικών υπηρεσιών Ας ελπίσουμε όμως ότι οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και των Εθνικών Υπηρεσιών δεν θα δημιουργήσουν ε, διαμάχες και κάποια διαφιλονικούμενα ζητήματα. Ε, στον ε, τομέα της αεροπλοείας μας είπαν ότι τα κατάφεραν πολύ καλά χωρίς να υπάρχουν ε, σοβαρά προβλήματα και θα πρέπει να ελέγξουμε αν αρκεί η νομοθεσία στον τομέα αυτό για να μπορέσει να ε, το καλύψει το θέμα. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο όμως ε, ε, να κατέβουμε σε μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειες από αυτό που προτείνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα αλληλένδετα ζητήματα με τα θέματα της διαλειτουργικότητα και άλλα θέματα και από και υπάρξει ασφάλεια δικαίου, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αρκετά θέματα και να συνεργαστούμε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Ρικέ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Ρόμπερτ Τζίλε για τη δουλειά του. Η άποψή μας είναι ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων θα πρέπει να αποτελεί το μοχλό ο οποίος ε, θα καθορίζει όλες τις ε, πτυχές ε, διαλειτουργικότητας και συνεργασίας στην Ευρώπη και γι' αυτό είμαστε υπέρ της ενιαίας σειρίδας σε αυτό το τομέα να είναι αρμόδιος οργανισμός για την πιστοποίηση όπως καθορίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης και το θέμα των ελέγχων κυρίως για το RTMS. Το πρόβλημα το οποίο ε, ε, αναφέρεται συχνά είναι τι γίνεται με τις εθνικές υπηρεσίες. Ε, θεωρούμε ότι υπάρχει τρόπος να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και των Εθνικών Αρχών, κυρίως για χώρες οι οποίες έχουν κάποιες ιδιωτηρότητες στις υποδομές τους, παραδείγματος χάρη τις Βαλτικές χώρες ή την Ισπανία ή ε, ε, όταν κάποια δίκτυα περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο. Ε, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, αλλά υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για να υπάρχει αντίστοιχη ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ε, στοιχείο ε, υπέρ της Ευρώπης, της σημαντικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το γεγονός για παράδειγμα ότι ε, το προσωπικό το οποίο βρίσκεται επί των ε, ε, σιδηροδρομικών οχημάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένο, θα πρέπει να διορθώνονται και κάποιες δευκρινήσεις για το τι έγινε και υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για την εσωτερική ε, των πραγμάτων. Και επίσης θα πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις στο δεύτερο κεφάλαιο τι γίνεται με την ε, ε, ευθύνη του οργανισμού και την ε, ανεξαρτησία του και επίσης θα πρέπει λίγο να δούμε και την ανθρώπινη αλλά και την οικονομική πτυχή. Διότι πολλά από αυτά τα καθήκοντα ναι μεν φαίνονται πολύ σημαντικά, αλλά οι μέσες προβλέψεις είναι μάλλον αβέβαιες, θα ήταν ε, ε, ρηψοκίνδυνο να αναθέσουμε καθήκοντα τόσο σημαντικά σε έναν οργανισμό ο οποίος δεν έχει κατάλληλο προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσει. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί ο χρόνος σε όλους τους ε, διαχειριστές ε, να μπορέσουν να προσαρμοστούν και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει και κάποιο συμβιβασμός αφενός ε, για το τι γίνεται με τις ε, προτινόμενες προθεσμίες. Κάποιοι προτείνουν ένα χρόνο, υπάρχουν τροπολογίες που προτείνουν από μηδενική διαφορά με μεταβατική περίοδο μέχρι περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε πόσο σημαντικές θα είναι οι αλλαγές και αν θα πρέπει να προσέξουμε ε, και τα μέσα και τις προθεσμίες και το πότε θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Γκρινιό για δύο λεπτά. Παρνιό, συγγνώμη, για δύο λεπτά. Ε, εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων που εδρεύει στη Βαλενσιέν της Γαλλίας και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα να απευθύνεται κάποιος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την πιστοποίηση, αλλά και στον Εθνικό Οργανισμό και αυτή η παρέκκληση θα πρέπει να αποτελέσει εξαίρεση, να είναι η μόνη περίπτωση στην οποία θα αποφασίζει κάποιο αν θα πρέπει να αποτανθεί στην Εθνική Υπηρεσία ή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Έχουμε προτείνει κάποιε τροπολογίε που θεωρούμε ότι βελτιώνουν τι διατάξει, διευκρινίζουν λίγο τα καθήκοντα και τι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και ε, τι αρμοδιότητες έχει αυτός ο οργανισμός ε, για την ανάκληση και την ε, ακύρωση αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο παρελθόν, τι γίνεται επίσης με τις ποινικέ ευθύνες του οργανισμού και του προσωπικού, τι γίνεται με την αβιβαία πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών, να βελτιώσουμε λίγο καλύτερα το γλωσσικό καθεστώς του οργανισμού και να υπάρξει και μια μεταβατική περίοδος όπως υπενθύμησε και ο συνάδελφος Ντομινίκ Ρικέ, ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να αυξήσει το δυναμικό του και τις δυνατότητές του για να έχει ταυτόχρονα και τους κατάλληλους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη για να διαχειριστεί το νέο του ρόλο ως υπεύθυνο για την σιδηροδρομική ασφάλεια. Αυτή η μεταβατική περίοδος θα μπορούσε ίσως να είναι αντίστοιχη με αυτήν που είχαμε ε, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ε, Ασφάλεια στην ε, Αεροπορία ε, και επομένως να έχουμε δύο στάδια, δύο χρόνια μεταφοράς και τριάμιση χρόνια για την ε, μεταβατική περίοδο στην οποία θα μπορούν ακόμα τα κράτη-μέλη να εκδίδουν τα προστοπικά και τις εγκρίσεις υπό την αίρεση του ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, ιδίω όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας και τη μη διάκριση για τις συγκεκριμένε αυτές άδειες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Ρόμπερτ για τη δουλειά που έκανε και τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους. Χαίρομαι που νομίζω ότι φτάνουμε κοντά σε μια λύση για κάποια θέματα, κυρίως για τις αυστηρές ε, προθεσμίες που αποτέλεσαν και στο παρελθόν ε, πρόβλημα και για το σύγκρουση συμφερόντων. Νομίζω ότι και εκεί έχουμε βρει κάποια λύση. Ένα ερώτημα για την Κομισιόν έχω σε σχέση με κάποιες προτάσεις που γίνονται στις τροπολογίες για τους ταχογράφους, για τους οδηγούς ε, τρένων. Για τις οδικές μεταφορές, εντάξει, είχαν υπάρξει κάποιε περιπτώσεις κατάχρησης, αλλά υπάρχει τέτοιο περιπτώσεις κατάχρησης στις συνδρομικές μεταφορές. Και για τις σιδηροδρομικές μεταφορές ο, ο, μπορεί να σταματήσει το τρένο ο οδηγός αν ο ταχογράφος είναι δεν, είναι, δεν δουλεύει σωστά, αλλά με τις καθυστερήσεις που θα υπάρξουν δεν θα γίνει. Επίσης, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις ε, για το θέμα αυτό, της επιλογής δηλαδή μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και της Εθνικής ε, Εταιρείας που ε, έχουμε να επιλέξουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε μακροπρόθεσμα να διατηρήσουμε μια τέτοια δυνατότητα. Εγώ δεν έχω βέβαια πρόβλημα να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος προς αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε μία τιμή για τους πάντες και μία λύση για όλους. Δεν γίνεται να χρεώνουμε την Deutsche Bahn το ίδιο που χρεώνουμε μια μικρή περιφερειακή εταιρεία που κάνει ένα δρομολόγιο 20 χιλιόμετρων. Είναι προφανές ότι κάποια μορφή προσαρμογή ανάλογα με τον χώρο χρήση θα πρέπει να υπάρξει. Έχουμε υποβάλει κάποιε τέτοιε τροπολογίε λοιπόν ε, με αυτόν τον όρο το area of use. Αλλά αν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο πρέπει να υπάρξει διαφορετικό κόστο ανάλογα με τον χώρο χρήση. Ε, είναι καλύτερα λοιπόν να υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γιατί αυτό έτσι θα πιέσει τις επιχειρήσεις, τις οδρομικές να δουν και πέρα από τα δικά του όρια και αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια με για τις βαλτικές χώρες εντάξει είναι ειδική κατάσταση, αλλά οι χώρες της βαλτικής θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα δικό του χώρο χρήση. χρήσης. Και θα έλεγα και κάτι για κάτι άλλο, αλλά το ξέχασα, οπότε θα σταματήσω εδώ. Κύριο Κράμερ, ναι, να ευχαριστήσω και εγώ τον Ρόμπερτ για την πολύ καλή συνεργασία και για τα θέματα που συζητήσαμε μαζί. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Μπορεί να μην είμαστε πάντα τη ίδια άποψη, αλλά προσπαθούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καλή. Για τι τροπολογίε τώρα. Η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό ω ενιαία θηρίδα ε, γίνεται αποδεκτό από, τους, ε, από πολλούς συναδρέφους. Ε, μιλήσαμε για, τον για, τους, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και του Εθνικού που επίση θα πρέπει να συνεργαστούν. Βεβαίω και οι περιφερειακέ και οι τοπικέ αρχέ κάνουν πολλή δουλειά, αλλά ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό θα έχει τον τελευταίο λόγο. Ε, τώρα για τα κοινωνικά θέματα βεβαίω τα υποστηρίζουμε, βεβαίω ε, μιλούμε για την ασφάλεια εδώ. Έχουμε υποβάλει σχετικέ τροπολογίε και μιλούμε για ε, ενίσχυση. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ καλά με αυτούς τους πίνακες που θα υπάρχουν, γιατί έτσι θα είναι πιο σαφή τα πράγματα. Ε, τώρα, για την διατύπωση, καλό θα ήταν να έχουμε μια ενιαία έτσι, ορολογία. Ε, αν τώρα υπάρξουν προβλήματα, ε, εντάξει, αυτό μπορούμε να το λύσουμε με τους... Ε, ε με όσους μιλούν την αγγλική ως μητρική. δεν υπάρχει τόσο τρομερό πρόβλημα πια. το σημαντικό είναι να έχουμε μία συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και των Εθνικών και γι' αυτό χαίρομαι που για την ασφάλεια, και τουλάχιστον για την ασφάλεια, ο γερμανικός οργανισμός ε, έκανε λίγο πίσω και δέχτηκε να έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός τον τελευταίο λόγο. Τώρα για τις ε, διάφορες αρμοδιότητες, ναι πρέπει να είναι σαφής, αλλά ε, όχι για πάρα πολλά χρόνια. Και το επόμενο βήμα είναι να δούμε τι θα γίνει με τις εξελίξεις στο Συμβούλιο να δούμε πώς θα προχωρήσουν και οι υπόλοιποι φάκελοι και για τη διαλειτουργικότητα. Νομίζω ότι θα βρούμε λύση εκεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε και στον κανονισμό για τον οργανισμό μια λύση. Αλλά επειδή είναι, ήταν πολύ καλό το κλίμα της συνεργασίας μας, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και πάλι ευχαριστώ τον Ρόμπερτ αλλά και την κυρία Μπιλβάου. Eh, Ο κύριος Κόλιτσεκ να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. <coughs> Καταρχά για το θέμα των δυνατοτήτων. Αν θέλουμε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός μετά από μια σύντομη μεταβατική περίοδο να μπορεί να κάνει άμεσα όλα τα τεχνικά τεστ, όλες τις τεχνικές δοκιμέ, ε, τι να πω, αυτό είναι παράλογο από, την, ε, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Πρέπει να ζητήσουμε να ορίσει τα πρότυπα και τα, τις δοκιμές να τις κάνουν οι, οι τοπικές αρχές. να γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Η ε, Ευρωπαϊκή Αρχή πρέπει να, να δει αν τα πρότυπα. Αυτό πρέπει να εξασφαλίσει, ότι θα γίνονται αμοιβαίω αποδεκτά τα σχετικά πιστοποιητικά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ε, βήμα προς τα εμπρός για τους σιδηροδρόμους. Και επίσης, Πρέπει να δούμε τα πρότυπα συντήρησης, ανεξάρτητα αν μιλούμε για την υποδομή ή για τα οχήματα. Και αυτό θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Και αν θέλουμε και αυτό να το κάνουμε και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προφανώς θα είναι τεράστια νίκη και για μας και για τις επόμενες γενιές. Πάμε στην τελευταία τώρα έκθεση του κυρίου Κόλιτσεκ. Για την ε, διευθέτηση των λογαριασμών. Τρία λεπτά στον κύριο Κόλιτσεκ και δύο στους ε, σκιώδεις. Κύριε Κόλιτσεκ, ευχαριστώ. Λοιπόν, για τη δική μου την έκθεση, ε, ήδη υπόθηκαν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ ενδιαφέρουσα. αλλά δεν ε, ενισχύει τους ε, σιδηροδρόμους. Αν ε, θέλουμε να, τους, να υποστηρίξουμε τους σιδηροδρόμους πρέπει να το πράξουμε υπεύθυνα και έναντι των υπολείπων τρόπων μεταφορών. Οι περισσότερες διατάξεις του 34-2012 θα ισχύουν μέχρι το 2015. Μάλλον θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το 2015. Το να αρθεί αυτό δεν είναι καλό. Αν τώρα η Κομισιόν λέει στην έκθεσή της ότι όλα είναι καλά, εγώ δεν είμαι απόλυτος πεπισμένος. Γιατί, γιατί όταν μιλάω με υπουργούς ε, μεταφορών, ή με κάποιον που δεν γνωρίζει απολύτως το τι γίνεται για το πώς έχει η κατάσταση, πάντα λένε ναι θα αρθούν αυτές οι διατάξεις. Αλλά αν μιλήσουμε με τους ε, εκπροσώπους των, ε, οργανώσεων σιδηροδρόμων, αυτοί πάντα λένε μην κάνετε τέτοιο πράγμα, μην, ας μην αρθούν αυτές οι ε, διατάξεις. Και τώρα πείτε μου, πιστεύετε ότι Καλύτερα γνωρίζει κάποιος υπουργό το τι γίνεται ή καλύτερα γνωρίζει ε, ένας εργαζόμενος στους ε, σιδηροδρόμους ή ένας που έχει άμεση σχέση και εμπειρία με τον κλάδο αυτό. Εγώ δούλευα σε μια τέτοια εταιρεία 23 χρόνια ε, και νομίζω ότι αυτός που εργάζεται και είναι η καθημερινή του δουλειά αυτή ξέρει πολύ περισσότερα από τον οποιοδήποτε υπουργό. Έχουμε το όριο του 2019 και μετά το 2015 λέει η Κομισιόν ότι θα τα αξιολογήσει όλα με μια έκθεση που θα λάβουμε το αργότερο 31 Δεκεμβρίου του 2017. Δείτε τι γίνεται με το... Δείτε τι έγινε με το Κώστα Κονκόρδια και το δυστύχημα. Μέχρι τώρα έκθεση δεν έχει υπάρξει. Οπότε νομίζω ότι μετά από δύο χρόνια από την ε, εκπνοή της προθεσμίας θα πρέπει να υπάρξει η σχετική έκθεση. Και όταν εκπνεύσει η οδηγία του 2012 θα πρέπει να υπάρξει από την Κομισιόν μια νέα μαθηματική πρόταση για να υπάρξουν τα ίδια, ίδιες διατάξεις για τους, για τις, ε, και για τις νέες εταιρείες τις υδροδρομικές, για όλες να, να υπάρχουν οι ίδιες προϋποθέσεις όλες οι εταιρείε που είναι στην αγορά σήμερα και δραστηριοποιούνται. Δεν θέλουμε να υπάρξει διακριτική μεταχείριση έναντι κανενό. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το μέγιστο, στο μέγιστο δυνατό βαθμό της διατάξης αυτής της, διατάξης, της, αυτής της ε, οδηγίας ε, προς όφελος των ε, ταξιδιωτών. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, για αυτή την πρόταση εξαίρεσης, εξαίρεσης θα ήθελα να συμφωνήσω με τον εισηγητή η εφαρμογή της οδηγίας για δημιουργία νέου ευρωπαϊκού συνδρομικού χώρου αναπόφευκτα θα αλλάξει το ρυθμιστικό τοπίο ε, στον τομέα αυτό και άρα δύσκολο είναι πρόωρο να ξεκαθαρίσουμε αν αυτό που προβλέπει ο κανονισμός για τις αποζημιώσεις πρέπει να εγκαταλειφθεί ως ιδέα και γι' αυτό, ιδέα, συγγνώμη, και γι' αυτό υιοθετούμε αυτή τη θέση και εξάλλου σε σχέση με την τοποθέτηση του εισηγητή θα έλεγα ότι σε αυτό το στάδιο, ε, στάδιο είναι καλύτερο να μην ορίσουμε η ημερομηνία γιατί θα ε, έπεται και η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ακούσαμε για το 2017. Αυτή η ενδιάμεση αξιολόγηση θα μας επιτρέψει να αποφασίσουμε αν ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να ε, καταργηθεί ή να τροποποιηθεί και γι' αυτό κατέθεσα διάφορες τροπολογίες εξυπηρετώντας αυτό το σκοπό. Ευχαριστούμε κύριο Σοντίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τις αμφιβολίες του εισηγητή του κυρίου Κόλιτσεκ και δεν θα πρέπει να διαφορούμε. Πρέπει όμως να σας πω ότι Εσκεμένα δεν παρουσίασα τροπολογίες στην πρόταση αυτή, διότι θεωρώ ότι είναι σωστή η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, η ανάγκη να βελτιώσουμε τον ε, ε, κανονισμό 1982 του 69 για την ε, διαθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Παρά τα όσα λέει ο εισηγητή, πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα κανονισμό ο οποίο ε, τέλο πάντων τα έχει φάει τα χρονάκια του και είναι πλέον παροχημένο. Όταν ο προπολογισμό των διαχειριστών των σιδηροδρομικών ε, ε, οργανισμών περιλαμβανόταν στον προπολογισμό του κράτους και έπρεπε το κράτος να εγγυηθεί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ε, τις ε, συντάξεις και τις ασφαλίσεις των υπαλλήλων ή να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες ε, απαιτήσει υποδομές, κυρίως για την υλοποίηση των διαφόρων διαδρόμων και περασμάτων. Ο κανονισμός αυτός ήταν εναρμονισμένος μεν, αλλά επέτρεπε σε 36 επιχειρήσεις μόνο να λαμβάνουν αποζημιώσεις. Σήμερα, υπό το φως της εναρμόνισης, είναι σαφές ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός είχε μεν κάποιο νόημα όταν οι ε, σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έπρεπε να προσέχουν μόνο τον ανταγωνισμό με άλλα μέσα μεταφοράς, όχι τον εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων διαχειριστών ε, της ίδιας υποδομής. Και επομένως, δεν είναι δυνατόν τη σήμερα ημέρα να γίνονται διακρίσεις. Και επίσης δεν είναι δυνατόν να γίνει επέκταση όπως θα ήθελε ο ε, πράσινος συνάδελφος για όλες τις επιχειρήσεις και θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την κατάσταση και να δεχτούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν ε, θέλει κάποιο άλλο το λόγο, γιατί δεν έχουμε όλου του εδώ. αλλιώς να ακούσουμε την Επιτροπή. Μάικλ. Ε, Έχω να σας αναφέρω την άποψη του συναδέλφου που συμφωνεί με την έκθεση του Κόλιτσεκ. Βεβαίως μιλά υπέρ της συνεργασίας και η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί μετά, δύο-τρία χρόνια μετά το άνοιγμα της αγοράς. Να μην αποφασίσουμε δηλαδή από τώρα και να μείνουν τα μέτρα ενισχύ. Ευχαριστώ Μάικολ. Ωραία. Κομισιόν. Τελευταία φορά σε αυτή την Επιτροπή. Θα σας δώσω 10 λεπτά για να μας εξηγήσετε την έκθεση. Βεβαίως δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσετε όλα αν δεν τα θέλετε, αλλά εμείς θα σας τα δώσουμε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι εξίσου αποτελεσματικός όσο και εσείς. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τους Βιλμπάου Κράμερ και Τσίλε για τις τρεις εκθέσεις σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Ε, είναι εξαιρετικές οι εκθέσεις, δείχνουν συνοχή στις θέσεις που προβάλλονται και από πολλές πλευρές βελτιώνουν και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι επίσης χρήσιμες οι προτάσεις ε, διότι υιοθετούν αυτή την έννοια της περιοχής χρήσης και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό κοινό έδαφος ε, για να εισέλθουμε στις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Ως προς τη συνοχή και την, ε, τους ορισμούς ε, σε αυτές τις εκθέσεις έχουμε υλικό στη διάθεσή σας. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια μονομένα ζητήματα που ε, ακούσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Το RTMS πρώτα απ' όλα είναι κάτι που αναφέρεται και στις τρεις εκθέσεις και είμαι ευγνώμων προς τους τρεις συγητές διότι συστήνουν όχι μόνο τα ίδια τα συστήματα RDMS για τα οχήματα αλλά και για τις υποδομές να καλύπτονται από τις αρμοδιότητες και τη διακυβέρνηση που θεσπίζονται βάσει αυτών των τριών εκθέσεων αλλά εξίσου σημαντικό είναι όπως είπε και ο Μάικλ Κράμερ διότι διευκολύνεται η μεταφορά στο νέο σύστημα τη migration που οδήγησε σε καταστροφικά μας είπα, τα αποτελέσματα δεν πήγαινα τόσο μακριά, αλλά τέλος πάντων μας οδήγησαν στο ρυθμό, στο ε, επίπεδο απογοήτευσης ε, με τη χρήση του RTMS στα δίκτυα. Αυτό δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά όπως είπε ο κύριος Κράμερ, για την ε, ανάπτυξη των προγραμμάτων RTMS, ε, το χαρακτηριστικό διαλειτουργικότητας, δεν καλύπτεται πάντοτε επαρκώς κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων και γι' αυτό και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός κρίνει ότι αυτό έχει την κέρια σημασία πλέον ούτως ώστε να θέσουμε ένα πλαίσιο για τους διαχειριστές υποδομών και για την εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων ε, του νέου κανονισμού. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που το τονίσατε και στις τρεις εκθέσεις. Δεύτερο σημείο κλειδί, οι πόροι. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες για τις ε, συναδέλφων και προτάσεις μέσα στις τρεις εκθέσεις για αυτό το ζήτημα. Ε, το μήτρο οχημάτων είναι ένα πιο συγκεκριμένο θέμα που θα μπορούσε να μας προσφέρει και μία λύση, η αρμοδιότητα εποπτείας των ελεγκτικών οργάνων, κάτι που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενισχύεται και εσείς με τις τροπολογίες που καταθέσατε. Καλωσορίζουμε αυτή την ιδέα. Βεβαίω αυτό έχει σημαντικότερες επιπτώσεις ως προς τους πόρους. Ο Ντομινίκ και διάφοροι άλλοι το επισήμαναν. Και όντω το ζήτημα είναι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Δημοσιονομική Αρχή θα σταθεί στο ύψος των ε, προκλήσεων ε, των συνομοθετών ως προς τον κύριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ε, και θα μας βοηθούσε αυτό να αποτιμήσουμε για τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια πρόταση σε ένα πιο προκεχωρημένο στάδιο της διαδικασίας. Και τελευταίο σημείο, το χρονοδιάγραμμα και η σταδιακή μεταφορά αρμοδιοτήτων, εκχώρηση αρμοδιοτήτων προ τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Εμείς προτείναμε αυτό να γίνει μετά τη λήξη της διετούς προθεσμίας για τη μεταφορά, για τις οδηγίες ασφάλειας και διαλειτουργικότητα ενώ έτσι η βιομηχανία θα έχει τις αποτελεσματικότερες μεθόδους που ε, ζητά, αλλά ταυτόχρονα με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα είναι χρονοβόρες, ε, ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός στο μεταξύ θα έρχεται σε επαφή με τις εθνικές αρμόδιες αρχές και γι' αυτό θέλω, όπως και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, να τονίσω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις νέες ευθύνες μετά το πέρας αυτής της μεταβατικής περίοδου για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Ε, ποιο είναι το σκεπτικό είναι η αναβαθμισμένη ποιότητα, καλύτερη διαλειτουργικότητα και ασφάλεια, αλλά αν τελικά το Κοινοβούλιο επιλέξει αυτή την άγουσα, θα δυσχεράνει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις, για το Συμβούλιο είχε προτείνει την πενταετή περίοδο για τη μεταφορά, πρέπει να το έχετε και αυτό κατά νου. Ε, όλα τα υπόλοιπα σχόλια μου είναι τεχνικού χαρακτήρα για τις τροπολογίες. Ο Μάικλ, ο Πίτερ Λίζη και εγώ και οι υπόλοιποι σκιώδεις θα τα δούμε μεταξύ μας, αν συμφωνείτε. Για την έκθεση Κόλιτσεκ, για τις ανταλλαγές, έχουμε κάνει μια αξιολόγηση της χρήσης και της χρησιμότητας ε, αυτού του ε, απαρχαιωμένου κανονισμού. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι πρόταση έχει προσθεμένη αξία και στις διάφορες κατηγορίες αυτού του κανονισμού έχουμε υποκατηγορίες που ήδη καλύπτονται και φαίνεται ότι Υπάρχει κείμενη νομοθεσία ή αναθεωρημένα νομοθετήματα που καλύπτουν τις διάφορες κατηγορίες και η πρόταση που εξετάζουμε τώρα δεν προσθέτει τίποτα σε σχέση με αυτά. Ε, αυτό σχετίζεται με το θυματολόγιο τη καλύτερη νομοθεσία και ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό προσπαθεί να κάνει. Δεν είναι εύκολο, ε, εύκολη άσκηση. Έχουμε βεβαίως ένα ιδανικό υποψήφιο για να το καταφέρουμε. Είναι ουδέτερη η αξιολόγηση που κάνουμε, όμως ε, το γραφειοκρατικό άχθος είναι η Ε, είμαστε στη διάθεση όλων των ε, εισηγητών ε, και του κύριου Κόλτσεκεν προκειμένου για να συζητήσουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων επί τόπου. αυτές οι ανησυχίες προκύπτουν εν μέρει από την άγνοια της κείμενης νομοθεσίας και άλλων υφιστάμενων διαδικασιών, οπότε μπορούμε να προσπαθήσουμε να καθησυχάσουμε τους φορείς ότι η κατάργηση αυτού του κανονισμού είναι και προς όφελός τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε θα ήθελα τώρα να σας ευχηθώ ότι καλύτερο στην επόμενη μετάθεσή σας εντό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να σας ευχαριστήσω για τα όσα κάνατε εδώ με την Επιτροπή Μεταφορών, τουλάχιστον για όσο διάστημα ήμουν εδώ εγώ στα ενία. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στην επόμενη μετάθεσή uh, σας. ευχαριστώ πολύ, Μπράιαν, και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους σας. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας ευχαριστήσω και εσάς προσωπικώς και να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη και όλο το προσωπικό για την εξαιρετική συνεργασία, την οποία είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια πλέον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Να δώσω απευθείας το λόγο στους εισηγητές. Ο κύριος Αλκαντράου δεν έχει τίποτα να πει. Ο Ντομινίκ έχει να πει τα περισσότερα του κυρίου Γκρός. Πολύ γρήγορα, ο Ματία Γκρός μας επισημαίνει ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει τους συναδέλφους για τη συνεισφορά του. Ε, να μας πει ότι συνειδητοποιεί φυσικά ότι θα πρέπει να καταλήξει σε συμβιβασμού και λέει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή η διάθεση ε, συμβιβασμού απευθύνεται και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εκεί και πέρα αυτό που έχει ως στόχο είναι η βελτίωση των υπηρεσιών και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μειώσουμε και τους κοινωνικούς όρους που έχουμε και επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να πω δύο λόγια και εγώ στον κύριο Πακέ, να το εκφράσω την χαρά μου και την εκτίμησή μου προς το πρόσωπό του και είναι κρίμα που φεύγεται. Η κυρία Μπιλμπάου θέλει να πει κάτι. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Πακέ και την ομάδα του για την εξαιρετική τους δουλειά και τη συνεργασία πάντα ήταν στη διάθεσή μας ε, και ήθελαν να συνεργαστούν τουλάχιστον με την Επιτροπή μας και με την υποφαινόμενη. Συνοψίζοντας να πω απλώς ότι χαίρομαι διότι τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει κάπως να προοδεύσουμε και να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Ε, θα υπάρξει μια κρεμότητα, να δούμε πώς θα γίνει η μετάβαση ε, μέσω στον τρόπο ώστε να υπάρχει κατάλληλη εναρμόνιση η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τους φραγμούς που αποτελούν ανάχωμα στη βελτίωση των σιδηροδρόμων και φυσικά ε, να δούμε τι στόχους ε, πρέπει να έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Ε, να πω ότι είμαι ικανοποιημένη διότι όλες οι τροπολογίες που υποβάλαμε που αναφέρονται στα άτομα με μειωμένη κοινωνικότητα και αναπηρία έγιναν δεκτές καθώς επίσης και την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό μητρό με κάποιες αποχρώσεις οι οποίες νομίζω θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Και όσον αφορά το θέμα των δικτύων, νομίζω ότι θα πρέπει να τα συζητήσουμε και τις ε, ε, προθεσμίες μετάβασης και μεταφοράς σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό που χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ. Σας ευχαριστούμε ε, για την αγαστή συνεργασία. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω προσωπικά και τον συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις, ε, διαφωνήσαμε συχνά για πολλά ζητήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ βεβαίως όταν έρχομαι κάθε, φορά, κάθε πρωί στη δουλειά, τον βλέπω πάνω στο ποδήλατό του εδώ δίπλα. Πάνε χρόνια λοιπόν που συνεργαζόμαστε και ε, θα ήθελα να τον ε, ευχαριστήσω, θα του δώσω δώρο και ένα βιβλίο. Τον καλό να έρθει και στο Βερολίνο για να του παρουσιάσω την κατάσταση εκεί σε πώς σας ευχαριστούμε. Τι θέλετε να προσθέσετε κάτι, ναι. κύριε Τσίλε, ναι. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον συνάδελφο. Είναι ιδιαίτερα επαγγελματίας και ήταν πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Νομίζω ότι για τα τεχνικά ζητήματα δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές, οπότε ας σκεφτούμε και αυτό το ενδεχόμενο να τα βρούμε σε πιο προσωπικό επίπεδο. Κύριε Κόλτσακ. Ε, ε, Θα ήθελα να δω και εγώ τον κύριο Πακέ στο ποδήλατό του. Όχι μόνο εδώ, στις Βρυξέλλες, αλλά και στο Βερολίνο και γιατί όχι στη δική μου την πόλη. Εγώ πιστεύω ότι μετά από κάθε ανταλλαγή απόψεων πρέπει να είναι κανείς συνετός να αξιολογεί την κατάσταση και να επιτρέψουμε σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου να διευθετήσουν τα ζητήματα με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Δεν είναι και χιλιάδες οι επιχειρήσεις ε, στον σιδηροδρομικό κλάδο, ενώ αυτές που ευθύνονται για την υποδομή και η πλειοψηφία παρέχει υπηρεσίες. Εκτιμώ ότι περίπου 40-50 επιχειρήσεις στην Ευρώπη διαχειρίζονται την υποδομή και άρα μπορούν να αποκομίσουν ωφέλη από αυτήν την ε, νέα πρόταση. Όμως η προθεσμία δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλη. Να συνεχίσουμε λοιπόν τις συζητήσεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο πρωταρχικός στόχος όλων μας είναι ο τομέας των σιδηροδρομικών μεταφορών να γίνει πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τους άλλους κλάδους και ενδεχομένως να τους βοηθήσει στην οικονομική τους ανάπτυξη. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τι προβλέπετε στις 26 Νοεμβρίου να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Πιέζονται οι συγητές και οι σκιώδεις σε μεγάλο βαθμό λοιπόν για να καταλήξουν ή δυνατόν σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις μέχρι τότε. θα συνεχίσουν οι συζητήσει και φαίνεται ότι για τον τεχνικό πυλώνα είναι σχετικά ξεκάθαρη συνενετική λύση που έχουμε βρει. PSO, και άνοιγμα της αγοράς είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Το μόνο μπορώ να κάνω εγώ και το απαιτεί ο ρόλος μου είναι να ενθαρρύνω όλους τους εμπλεκόμενους, εισηγητές και σκιώδες να δείξουν καλή θέληση γιατί μόνο έτσι θα τα βγάλουμε πέρα. Ευχαριστώ επίσης ε, για την πειθαρχία που δείξατε. Τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα και ε, νιώθω και ήσυχο ότι ακούστηκαν όλες οι φωνές κατά τη διάρκεια της συζήτησης και έχουμε μια ε, καλή θέση. 26 Νοεμβρίου λοιπόν ψηφοφορία στην Τραν. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα. Θα σας πω μόνο ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου, στις 3 Δευτέρα, εδώ στις Βρυξέλλες. Θα σας δω τότε και θα αρχίσουμε, αν μπορέσει κάποιος να βρει το ματιό για, για μένα, να αρχίσουμε κατευθείαν τη συνάντηση συντονιστών. Α, δεν θα έρθει, καλά να αρχίσουμε τότε. Πεντάλεπτη διακοπή για να αρχίσει μετά η συνεδρία των συντονιστών.